Okay, colleagues. Η, προ... Πρόεδρος, ευχαριστώ που ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι και είπαμε να επενθυμίσουμε προς όλους τους συναδέλφους και το προσωπικό μας ότι πάντα το απόγευμα θα αρχίζουμε τρίτες και τετάρτες στις 2.30 ώρα το απόγευμα. Και όχι στις 3 ώρα. Με μεγάλη μας ε, ευχαρίστηση θα ακούσουμε την ε, Καταρίνα Ζαχαρίεβα που είναι η, υφυπουργός για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και την ε, παιδεία στην Βουλγαρία και θα μας πει τι γίνεται όσον αφορά την προσέγγιση της Προεδρίας για ζητήματα ε, ανθρωπιστικά και ασχολείται και με ε, την εξωτερική πολιτική της χώρας επίσης, προσθέτει πρόεδρος, οπότε θα πρέπει να σας πούμε ότι είχαμε την εντύπωση και οι συντονιστές ότι η Βουλγαρική Προεδρία παίρνει πολύ στα σοβαρά την πολιτική ανάπτυξης. Οπότε με μεγάλη μας ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε και ξέρετε από τότε που ανέβα πρώτα στην Επιτροπής πάντοτε λέγαμε ότι είναι τόση η παγκοσμία κρίση ότι χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια. Η μία κρίση μετά την άλλη συμβαίνει. Οπότε συνάδελφοι ε, και τα κακά μαντάτα είναι ότι στο Αφγανιστάν, στην Καμπούλ, τα γραφεία του Save the Children πέσαν τρομοκρατική επίθεση. Ε, είχαμε ε, απώλειες θανάτους από πλευράς του προσωπικού, δεν ξέρουμε ακόμα τις λεπτομέρειες. Και να, από εδώ καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνη είναι η δουλειά όσων ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια, πόσες δυσκολίες έχουν να αντιμετωπίσουν. Κύριε Υπουργέ, περιμένουμε πώς και πώς να σας ε, ακούσουμε. Ε, η συγκυρία είναι τέτοια που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ανθρωπιστική βοήθεια και έχετε τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διακεκριμένοι κύριοι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, δυστυχώς αυτά που μόλις είπατε ισχύουν. Και στην εισαγωγή μου θα αναφερθώ και σε ορισμένες άλλες νέες κρίσεις, καταστάσεις κρίσεων που προέκυψαν ε, μετά την ε, παρουσίαση της ε, Εστονικής Προεδρίας για αυτό το θέμα. Αυτό που συνέβη σήμερα στο Αφγανιστάν καταδεικνύει ότι δυστυχώς υπάρχουν πολλές επιθέσεις κατά των προσπαθειών που κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις ανθρωπιστικές κρίσει. και ορισμένε δυστυχώς είναι και από κυβερνήσεις. Πρέπει να το ξεχνάμε, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πρώτη μα προτεραιότητα πρέπει να είναι η συζήτηση για αυτό το θέμα και να εμείνουμε στην τήρηση των αρχών και το σεβασμό της ε, διεθνούς ανθρωπιστικής προσπάθειας. Και να ξεκινήσω την ομιλία μου με ορισμένα στοιχεία. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το 2018 τώρα, έχουμε πάνω με 145 εκατομμύρια άτομα που είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον κόσμο. Ε, τα 105 εκατομμύρια λαμβάνουν κάποια μορφή βοήθεια. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η βοήθεια που λαμβάνουν περισσότερο από αυτούς είναι επαρκής. Ανεξάρτητα από το συνεχώς αυξανόμενο ποσό της βοήθειας που παρέχει η διεθνής κοινότητα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα κενό χρηματοδότησης περίπου 25 δις δολαρίων μόνο για φέτος. Να σα δώσω μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα από συγκεκριμένε χώρε Στη Συρία. Μόνο στη Συρία υπάρχουν 13 εκατομμύρια σε κατάσταση ανάγκης. 2 εκατομμύρια από αυτά δεν λαμβάνουν καμία ανθρωπιστική βοήθεια. Στην Ιεμένη υπάρχουν 11 εκατομμύρια. Στην περιοχή Ρακίν της Μιανμάρ το 1 τρίτο των παιδιών υποφέρουν από υποσυτισμό. 60% του πληθυσμού της Λιβύης ε, χρειάζεται επιστηστική βοήθεια. Στο Νότιο Σουδάν έχουμε 2 εκατομμύρια εσωτερικά μετατοπισμένα άτομα. Στη, στο Κονγκό ο αριθμός είναι πάνω από 4 εκατομμύρια των εσωτερικά μετατοπισμένων. Και δεν θα σας πω και άλλα στοιχεία γιατί αν συνεχίσω δυστυχώς δεν θα μείνει καθόλου χρόνος για να αναφερθώ σε άλλα θέματα. Η Βουλγαρία καθώς και άλλα κράτη-μέλη διαπίστωσε την τρομερή επίπτωση του σημερινού ψηλού επίπεδου σειράξεων στον κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες μετατοπισμένα άτομα έχουν περάσει από τα σύνορά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται της συλλογική απαντήσεως του πλανήτη μας στις ανθρωπιστικές ε, ανάγκες. Ναι, βέβαια δεν έχουμε απεριόριστους πόρους, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε ανθρωπογενείς καταστροφές και σε θεομηνίες. Πρέπει να επιδιώξουμε να αντιμετωπίσουμε τις ρίζες των προβλημάτων. Διάφορες από τις ε, υπάρχουσες σειράξεις, ιδιαίτερα στην Αφρική, έχουν επιδεινωθεί λόγω της ε, ανομβρίας και των σειράξεων για την ε, μειωμένη πρόσβαση στην καλλιεργήσιμη γη και το νερό που χρειάζεται για τη γεωργία. Έτσι, για παράδειγμα, η σύγκρουση στο Νταρφούρ μπορεί να περιγραφεί ω η πρώτη σύραξη που προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή. Μερικέ από τι ε, πιο μακροχρόνιε σειράξει στον κόσμο είναι σε χώρε που είναι όλο και πιο άγονε, όπω το Νότιο Σουδάν, το Τσάντ και το Μαλί. Σύμφωνα με το δίκτυο για την ε, ε, ευπάθεια για την κλιματική αλλαγή, από τις 186 ε, χώρες το Τσάντ είναι πιο ευπαθής, η πιο ευάλωτη. Θεωρούμε ότι αν είναι, η απάντηση είναι μια, ένα συνδυασμό της μεταρρύθμιση του διεθνού Ανθρωπιστικού Συστήματος επιπλέον πόρη και ε, συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα και επίσης να υπάρξει περισσότερη χρήση του νέου ε, πλαισίου αντοχής της Ένωσης για να επιληθούν και να προληφθούν οι ε, σειράξεις. Πριν συνεχίσω θέλω να αποτίσω φοροτιμή στην εξαίρετη εργασία που έκαναν οι προκατοχοί μας, η Μάλτα και η Εστονία, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Και οι δύο χώρες βοήθησαν να, αντιμετωπιστούν, να εντοπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και να υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδος για να υπάρξει μια ευρεία συμφωνία για την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάπτυξη και για να υπάρχει νέα προσέγγιση για την ε, αντοχή. Βλέπουμε ότι δημιουργείται μια νέα στρατηγική. Σε μια συνάντηση τη Επιτροπής σας πριν από μερικού μήνε, ο, ο στονός συνάδελφος ε, Υπουργός Βεν Μίξερ ανέφερε ότι το πάνελ υψηλού επίπεδου για την ανθρωπιστική χρηματοδότηση των ΗΕ εντόπισε ότι υπήρχε ένα κενό χρηματοδότηση 15 δις δολαρίων για την παγκόσμια ανθρωπιστική δράση. Έχει υπάρξει ε, περιορισμένη πρόοδος έκτοτε, και οι ανάγκε στην, στην Ιεμένη, τον Νότιο Σουδάν, τη Σομαλία και τη Βορειοανατολική Νιγηρία εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Και επιπλέον ε, δημιουργήθηκαν και νέα προβλήματα σε άλλες περιφέρειες, ιδιαίτερα η μετατόπιση της κοινότητας των Ροχίνγκια, που είναι άλλη μια ανθρωπιστική κρίση που δημιουργήθηκε λόγω σειράξεω. Η παγκόσμια στρατηγική τη Ένωση για κοινή δράση και για να μην γίνονται οι ευαίσθητε καταστάσει ανθρωπιστικέ καταστροφές είναι το νέο μας όργανο. Θέλουμε να υπάρξει όλο και καλύτερα και πιο καλά συντονισμένη χρήση των ε, ανθρωπιστικών και διπλωματικών δυνατοτήτων της Ένωσης για να αντιμετωπίζονται τα αίτια των σειράξεων. Πρέπει να συζητήσουμε μαζί τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά για να αυξηθεί η συνοχή, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ε, κοινών μας ενεργειών. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια που εκφράζει τη δέσμευση της Ευρώπης να βοηθήσουμε τους πολίτες παντού στον κόσμο. Η Παγκόσμια Ανθρωπιστική Συνάντηση Κορυφής του 2016 στην Κωνσταντινούπολη κατέληξε σε μια σειρά από δεσμεύσεις από διάφορους ε, συμμετέχοντες και τα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής δημιουργούν ένα συνεπές πλαίσιο για τη σωστή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ε, τα πορίσματα αυτά και βασιζόμενοι στην εργασία των προηγουμένων προεδριών, η Βουλγαρική Προεδρία θα συνεχίσει να προωθεί συζητήσεις για την πρόοδο εφαρμογής αυτών των δεσμεύσεων και πρωτοβουλειών. Ιδιαίτερα θα ασχοληθούμε με την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και με τη μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος στην ε, διαδικασία ε, εφαρμογής των πορισμάτων τη Κορυφή, Η Ισπανία, Γαλλία, η Ιταλία και Πορτογαλία έχει ήδη ξεκινήσει μια σημαντική συζήτηση με ορισμένε ιδέε με μια πιο, για μια πιο συστηματική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι κρίσει ιδιαίτερα οι ξεχασμένε κρίσει. Η Προεδρία μα θα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να οικοδομήσει περαιτέρω με βάση αυτέ τι ιδέε και να διερευνήσει εναλλακτικέ λύσει για να δούμε πώ επιτηρούμε και διαχειριζόμεθα την αντίδρασή μα και στι ανθρωπογενεί κρίσει και στι θεομηνίε θα εξετάσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ε, διαδικασίας μεταξύ κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ανταλλαγή πληροφοριών για τον προγραμματισμό της αντιμετώπισης των κρίσεων. Θέλουμε να έχουμε συλλογική θέση για κάθε κρίση και έτσι θα καλύψουμε τις πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και μαζί με άλλους δωρητές που συντονιστούμε. Θέλουμε επίσης να υποστηρίξουμε και να τονίσουμε το ότι ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση για αυτή την έκκληση προς δράση για την προστασία από έμφυλη βία σε περίπτωση ε, ε, έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά πώς μπορούμε να κάνουμε βήματα να καταπολεμήσουμε ε, σεξουαλική βία και έμφυλη βία εντός των συζητήσεων επί συγκεκριμένων ανθρωπιστικών κρίσεων. Σχετικά με αυτό θα πρέπει να θεωρήσουμε, εξετάσουμε το δεκόμενο λήψεως πολιτικών μέτρων πέρα από την παροχή κάποιων να ληφθούν πρακτικά μέτρα πέρα από την ε, παροχή συμβουλών και παρενέσεων. Θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις, παραδείγματο χάρη, πώς ίδια προγράμματα και διαδικασίε μπορεί να προστατεύσουν γυναίκες, κορίτσια, ε, αγόρια και άντρε από τέτοια βία σε έκτακτες ε, καταστάσεις. Θα πρέπει να έχουμε πολιτικές συστήματα και μηχανισμούς ούτω ώστε να μειωθεί η έμφυλη βία και ο κίνδυνο αυτή τη βία, κυρίω να υπάρχει μείωση του κινδύνου κατά γυναικών και κοριτσιών και να παρέχουμε ασφαλεί υπηρεσίε εκείνου που επηρεάζονται από την έμφυλη βία. Μία από τις ανησυχητικέ συνέπειες της ε, παρούσης ανθρωπιστικής καταστάσεως στον κόσμο είναι η χαμένη γενιά των παιδιών που μεγαλώνουν σε στρατόπεδα προσφύγων σε καταβλισμού προσφύγων, από εκεί που του αρνούνται το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή παιδεία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε να, παρασχε... να δημιουργηθεί ένα αίσθημα κανονικότητα και να του δώσουμε ελπίδα και μια ευκαιρία να γίνουν παραγωγικοί πολίτε. Δεόντω λοιπόν η Βουλγαρία θα φροντίσει να παρέχεται ποιοτική εκπαίδευση σε ανθρωπιστικές έκτακτες ε, καταστάσεις και αυτό θα μπορούσε να μειώσει ε, τα επικίνδυνα κενά που διαπιστώνονται στην εκπαίδευση των παιδιών. Η παιδεία είναι θεμελιώδες για την ανθρώπινη, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και βασικό στοιχείο για να επιτευχθεί μια βιώσιμη ειρήνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι επιστημιστικές κρίσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο επί των πληττωμένων πληθυσμών και εκατομμύρια άνθρωποι διατρέχουν κινδύνους. Η Βουλγαρική Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται προς μια επαρκή συλλογική απάντηση, ούτως ώστε να αποφευθεί και να μειωθεί η πείνα ε, και η κακή διατροφή. Ε, ανέφερα ε, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο σχετικά με αυτά που συνέβησαν στο Αφγανιστάν, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό σαν θέμα και όλοι μας θα πρέπει να το θυμόμαστε και δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να το θέτουμε σε όλα τα μηνύματα που αποστέλουμε στους εταίρους μας να πούμε ότι είναι απαράδεκτο το να παραβιάζεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό ιδιαίτερα ενώπιον αυτή τη Επιτροπή, διότι το Ευρωκοινοβούλιο με συνέπεια ηγείται, ζητώντα η Ευρώπη να γίνει ε, ένα εταίρο γενναιόδωρο για ανθρωπιστικά θέματα και ανθρωπιστικά θέματα για τι κυβερνήσει και του λαού που χρειάζονται βοήθεια. Μπορείτε να βασιστείτε στην Βουλγαρική Προεδρία. Είστε βέβαιοι ότι θα επικεντρωθούμε επί πρακτικών δράσεων οι οποίε θα μπορούσαν να δώσουν ανθρωπιστικέ απαντήσει που είναι αποτελεσματικότερε και αποδοτικότερε. Προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σα του επόμενου μήνε και είμαι έτοιμη να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας και να ακούσω τυχόν προτάσεις και να ακούσω και τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ήδη πολύ συναδελφοί έχουν ζητήσει τον λόγο και τώρα ακόμα περισσότερο επομένως ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτό το οποίο είπατε. Συνήθως Πρώτος είναι ο κύριος Γκερέρο γιατί είναι ο μόνιμος συγχητής μας αλλά ο κύριος Βέντα από το ΕΛΚ ζήτησε να μιλήσει πρώτο. γιατί έχει υποχρέωση να πάει σε έναν τριμερή διάλογο. Ναι, ναι, πρόεδρε. Εντάξει, εντάξει, αφού δεν ενοχλεί το κύριο Γκερέρο οι άλλοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε για την εισήγησή σας, για τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας και με χαρά μου βλέπω ότι οι ανθρωπιστικές προτεραιότητες καλύπτουν και το θέμα της ε, κρίσης, της αντοχής και ανθεκτικότητας και οπότε βλέπουμε ότι οι χώρες εκείνες θα πρέπει να μην εξαρτώνται από εξωτερική βοήθεια για να επιλύσουν και να βγουν από τις κρίσεις που τις ε, χτυπάνε. Άρα αυτή η υπόθεση της ε, ανθεκτικότητας είναι πολύ σημαντική. Τώρα δούμε όσον αφορά αυτό τον ε, ανθρωπιστικό δεσμό, νέξους. Είναι και αυτό προτεραιότητά σας και σας ερωτώ. Πώς θα εξασφαλίσετε μια συνέχεια το να μην Έχουμε επικάλυψη δράσεων από τους εμπλεκομένους στα ανθρωπιστικά. Έτσι θα έχουμε και αποτελεσματικότητα. Και κάτι άλλο. Σημαντικό είναι η προεδρία σας όπως τονίσατε να κάνετε για την ανθρωπιστική κρίση ό,τι μπορείτε το οποίο θα αναβαθμίσει την αξιοπιστία της Ένωσης. Οπότε και σας ερωτώ. Για τις λεγόμενες ξεχασμένες κρίσεις έχετε κάποιο κατάλογο προτεραιοτήτων αναπεριφέρεια, περιοχή ή χώρα. και Γερέρο. Ναι, ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε, αλλά σας ευχαριστούμε και για το πρόγραμμα της Βουλγαρικής Προεδρίας. Θεωρώ ότι είναι ολοκληρωμένο ότι είναι πλούσιο σε ύλη γιατί τώρα για πρώτη φορά μια χώρα η δική σας χώρα λαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό δεν μπορεί παρά να προκαλεί ένα γενικευμένο αίσθημα εφορίας στην ε, χώρα σας. Ε, άρα έχετε ιδιαίτερο δυναμισμό σε σχέση με άλλες χώρες που έχουν αλλάξει την Προεδρία περισσότερες φορές οπότε εκεί δεν έχουμε τόση όρεξη και ξέρετε εδώ και πολύ καιρό αναλάβαμε για πρώτη φορά την Προεδρία όπως ξέρετε και θυμάμαι πολύ καλά αυτή την αισιοδοξία που είχαμε και μακάρι να κτηγήσεις μια αισιοδοξία το επόμενο εξάμεινο και να σημειώσουν πρώτα Τώρα Αναφερθήκατε βέβαια στο θέμα της ανθρωπικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο και όπως ξέρουμε καλά εδώ στην Επιτροπή μας. Όμως, εκτός αυτού του κοινοβουλίου, δεν νομίζω ότι έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος το ότι αυτή η παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση δεν είναι κάτι που σοβεί μόνο στην ε, Συρία, ούτε είναι μόνο θέμα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, Συρία. Ας πούμε στο Κονγκό, στο κυρίες της Αφρικής, σε διάφορα μέρη στην Ασία ή και Λατινική Αμερική και σε άλλες υπήρους. Έχουμε εκατομμύρια που κινδυνεύει η ζωή τους αυτή τη στιγμή γιατί τους λείπουν τα πιο σημαντικά, τα πιο στοιχειώδη το φαγητό για να επιβιώσουν. Οπότε τι θα κάνουμε με αυτές τις ξεχασμένες κρίσεις. Θα πρέπει τα κρατημέλη να ασχοληθούν και πάλι με αυτό. Αλλά βέβαια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την Προεδρία σας. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτές οι κρίσεις που δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις στα εσωτερικά των κρατών μελών της Ένωσης ε, παραμένουν παρόλα αυτά πολύ σημαντικές, πολύ έντονες ανθρωπιστικές κρίσεις Οπότε η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο γενικά προσπαθεί να αξιολογήσει πώς έχουν αποδώσει οι διάφοροι μηχανισμοί της ανθρωπιστικής δράσης, της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Οπότε τις αμέσως εβδομάδες θα προβούμε σε αυτή τη σφαιρική αξιολόγηση μαζί με την ΕΚΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα, για το τι γίνεται, πώς θα πάμε με την ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε και το Συμβούλιο Προεδρία σα θα εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία της αξιολόγησής μας και της Επιτροπής. Για να δούμε πόσο επιδέχονται βελτίωση όσα δεν πάνε τόσο καλά. Επίσης, μας ε, επισημάνεται ότι ένας από του στόχους ε, της μια Προεδρία μετά την άλλη είναι, όταν έρχονται εδώ να επισκεφθούν το Κοινοβούλιο, είναι να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις της συνάντησης κορυφής της Κωνσταντινούπολης του 16. Είχαμε στείλει αντιπροσωπεία σε αυτή την συνάντηση κορυφής και ο υποφαινόμενος είχα συμμετάσχει και ξέρουμε ότι δόθηκαν πολλές υποσχέσεις, πολλές δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Το λέγαμε το μεγάλο παζάρι, μεγάλη ευκαιρία, αλλά ίσως δεν είναι και τόσο δόκιμος αυτός ο όρος. Θα έπρεπε κάπως αλλιώς να το πούμε, κάτι πιο αλληλέγγυο. Θα έπρεπε να μην έχουμε έτσι υιοθετήσει έναν όρο, μια έκφραση που θυμίζει το παζάρι, το πάρε Οπότε και εμείς ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά θα προβεί σε κάποια παρουσίαση δεσμεύσεων θα ανατρέξει σε εκείνες τις υποσχέσεις της ανθρωπιστικής συνάντησης κορυφής και αυτή η αξιολόγηση θα αγγίξει τα κρατη μέσω των συναντήσεων του Συμβουλίου τώρα όσον αφορά το μέλλον. Κατάλαβα πόσα είπατε, πώς και εσείς ενδιαφέρεστε όπως εμείς ότι ο μηχανισμός της ανθρωπικής βοήθειας παραμένει μοναδικός στα πλαίσια των μηχανισμών δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί διέπεται από τις αρχές της ανθρωπικής βοήθειας και του ανθρωπιστικού δικαίου στο οποίο αναφερθήκατε πάνω από μία φορά στην ομιλία σας οπότε θεωρούμε ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν σε σίγουρο δρόμο. Θα πάμε και στο δήλωση του Μαΐου, στην πρόταση του Μαΐου, οπότε και εσείς θα πρέπει να τοποθετηθείτε σε σχέση με αυτή την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια που βέβαια τότε σχεδόν θα έχετε ολοκληρώσει τη διαδρομή της ε, Προεδρίας σας. Αλλά θα είναι σωστό να τα έχετε ήδη πει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτω ώστε την πρόταση αυτή να την αξιοποιήσετε τώρα όσον αφορά την ε, παιδεία για τα θέματα των δύο φίλων έχουμε τοποθετηθεί εμείς επανειλημμένως και στο μήκος κύματος στο οποίο κινηθήκατε κι εσείς αλλά να σταθώ σε κάτι συγκεκριμένο ε, βέβαια και είναι βασικό να φροντίζουμε για την παιδεία των ανηλίκων, των παιδιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν φύγει από κάποια κατάσταση δηλαδή που είναι πρόσφυγες ε, ή που είναι σε προβληματικές ε, χώρες όπως Τουρκία ή Λίβανο, εκεί που ε, εισραίουν εκατομμύρια ανηλίκων. Οπότε θα πρέπει να δούμε τους μηχανισμούς ανθρωπικής βοήθειας πώς μπορούμε να πλαισιώσουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή τα παιδιά πρόσφυγες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ακόμα δεν έχουν χαρακτηριστεί πρόσφυγες αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες ούτως ώστε να ενταχθούν στα σύστηματα εκπαίδευση των κρατών μελών σε πολλά κράτη-μέλη έχουν να εντάξουν στα σχολεία μέσα σε τρει μήνε από την είσοδό του αυτά τα παιδιά και μην έχουν χαρακτηριστεί πρόσφυγε. Και εγώ ξέρετε προεδρεύω σε κάποιο θεσμικό όργανο όπου στη χώρα μας δεν τηρείται αυτό, αυτό το τρίμηνο ένταξη στο σχολείο. Ούτε βοηθούμε αυτό τα παιδιά ιδιαίτερα όταν ε, πρέπει να μάθουν τη γλώσσα ή όταν θα πρέπει να ε, ανακτήσουν την, την ύλη του σχολείου που ε, έχουν χάσει επειδή έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους. Αν με ακριβώς έχουν χρόνο και οι άλλοι συνάδελφοι. Αλλά να σας πω εντάχει τα εξής επιπλέον. Πρώτα πρώτα. Σε λίγες εβδομάδες ή μήνες θα έχουμε τη δεύτερη διάσκεψη για την Συρία. Θα συγκληθεί από την κυρία Μογκερίνη και θα σας ζητούσα να εξωθήσετε τα κράτη-μέλη ως Προεδρία να ασχοληθούν δραστήρια με την ε, διάσκεψη αυτή για τη Συρία. Και κατά κλείδι, να δούμε κάτι που είπατε στο τέλος της ομιλίας σας. Μας μιλήσατε για το ότι χρειάζεται να προστατεύσουμε τους εμπλεκόμενους στα ανθρωπιστικά. Ε, είδατε τι έγινε με αυτή την επίθεση στο Save the Children και βλέπουμε ότι αυτό είναι κάτι τραγικό το οποίο συνέχεια γίνεται στους ε, πολέμους. Ομπαρδίζουν νοσοκομεία, σχολεία. Ε, θα πρέπει να αντιδράσουμε. Να αντιδράσουμε δυναμικά σε πολιτικό επίπεδο. Και οι κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα να προβάλλουν, να αναδείξουν, να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ρισκάρουν τη ζωή τους για να σώσουν τους ε, υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ Ενρίκε λέει η πρόεδρος και το λόγο στην κυρία Χόιποβα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά θέλω να υπερβώ αυτό το πλαίσιο. Στο πρόγραμμα εργασιών της Προεδρίας ε, αναφέρεται ορισμένα θέματα αναπτυξιακής πολιτικής. Θα ήθελα να κάνω ορισμένες ερωτήσεις για την επιστηστική ασφάλεια και τη γεωργία που συνδέονται πάρα πολύ με την ανθρωπιστική βοήθεια. γιατί πολλές φορές ε, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι παροχή επιστηστικής βοήθειας. Λοιπόν, για την ε, επιστηστική ασφάλεια. Κάθε δύο χρόνια ε, υποβάλλεται μία έκθεση πρόοδου από την Επιτροπή για το θέμα αυτό. Στην έκθεση αυτή υπάρχει μία επισκόπηση της ανα πάσα κατάστασης και Επίσης ε, αξιολογείται εάν η Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, τηρούν τις υποσχέσεις τους ή δεν τις τηρούν και σε τι βαθμό δεν τις τηρούν. Προβλέπετε το καλοκαίρι αυτή η έκθεση αυτή κατά την Προεδρία σας. Και κατόπιν θα υπάρξουν και συμπεράσματα του Συμβουλίου επ' αυτής της εκθέσεως. Όταν θα ασχοληθεί η ομάδα εργασίας ΔΕΦΚΟ με αυτό, Ελπίζω να μην ασχοληθούν μόνο με τις παλιές υποχρεώσεις για επιστηστική βοήθεια, αλλά να ασχοληθούν και με τις νέες υποχρεώσεις που έχουμε τώρα βάσω, βάση της νέας συνενέσεως που έχει επιτευχθεί. Θα ήθελα να υπάρξουν συμπεράσματα του Συμβουλίου που να βασίζονται και στις νέες αυτές υποχρεώσεις. Δεύτερη ερώτηση. Που και αυτή περιγράφεται στη συνένεση. Η Ένωση και τα κρατη τονίζουν ότι η βιώσιμη γεωργία και ιδιαίτερα η αγροοικολογία πρέπει να προωθηθούν. Θα ήταν πολύ ευχάριστο εάν το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του θα μπορούσε να αναφερθεί σε αυτές τις νέες υποχρώσεις που προκύπτουν από τη συνένεση και ιδιαίτερα λόγω του Διεθνούς Συμποσίου που θα διοργανώσει ο ΦΑΟ τον Απρίλιο για την αγροοικολογία. Υποθέτω ότι θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι αυτό το συμπόσιο που εγγράφεται σε αυτή την εντελώ νέα συνένεση θα ήταν η σωστή ευκαιρία για να προωθήσουμε την αγροοικολογία, να της δώσουμε μια νέα όθηση Και αγροοικολογία είναι ούτως, ούτως ή άλλως ο τίτλος αυτής της ε, λοιπόν, η Προεδρία σας να υποστηρίξει αυτή την εκδήλωση. Γιατί έτσι μπορεί να υπάρξει η αναγκαία αντοχή που λέμε. Ούτως ώστε όταν προκύψουν θεομηνίες, ξηρασίες, πλημμύρες να υπάρχει πολύ περισσότερη ανθεκτικότητα της οικονομίας, να είναι καλύτερα προετοιμασμένη η παραγωγή τροφίμων. Είδαμε τι έγινε με την ΑΕΤ, τι συνέβη. Οι περιοχές που ήταν πιο πολύ προσαρμοσμένες σε αυτήν την αγροοικολογία συνήλθαν πολύ ταχύτερα από τις άλλες περιοχές. Και αυτό σε τελευταία ανάλυση είναι μια προληπτική πολιτική που θα αντικαταστήσει την ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια εκ των υστέρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μυρίκ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, καταρχάς σας ευχαριστώ που ήρθατε να παρουσιάσετε στην Επιτροπή μας τις προτεραιότητες που καθορίζει η Προεδρία της χώρας σας όσον αφορά τα ανθρωπιστικά θέματα και την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Να επιστήσω προσοχή σας αν επιτρέπετε σε ένα σημείο που θεωρώ σημαντικό Πιστεύω ότι η ανθρωπιστική δράση θα πρέπει να συμπεραβάνει συγκεκριμένε και πραγματιστικέ στοιχείε. Η χώρα σα, κυρία Υπουργέ, ανακοίνωσε ότι θέλει να ζητήσει να βοηθηθούν τα εκτοπιστέντα άτομα στον κόσμο, οι πρόσφυγε, οι μετανάστε, με προέλευση ε, περιοχών σε κίνδυνο ή εμπόλεμε περιοχέ. Εγώ πήγα στο Ερμπίλ, στο Κουρδιστάν του Ιράκ και είδα το, το εκτοπισμένο πληθυσμό. Πήγα και στην Αφρική επανειλημμένα Πάντα ίδιες ανάγκες, οι θεμελιώδεις υπάρχουν και ζητούν βοήθεια αυτοί οι πληθυσμοί. Να μπορούν να ζουν ειρηνικά στη χώρα καταγωγής τους, να ανθίσει εκεί η ζωή τους και να αναπτυχθούν με τις χώρες τους. Η υποδοχή των προσφύγων κατά χιλιάδες στην Ευρώπη δεν μπορεί να ειδωθεί σε μια μακροπρόθεσμη αποτελεσματική λύση η ανθρωπιστική δράση σε αυτές τις περιοχές του κόσμου. Είναι θεμελιώδου σημασία, είναι καθήκον μας να συνεχιστεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η συνεχής έκκληση να πέσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα και να μπορούν να μπουν ολόκληροι πληθυσμοί που εκριζώνονται από τις περιοχές τους και χωρίς να έχουν προοπτική για το μέλλον σε μια εντελώς ξένη περιοχή είναι σε πλήρη αντίφαση με τους στόχους της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Το ερώτημά μου. Η Βουλγαρική Προεδρία θα φροντίσει ούτως ώστε η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να επικεντρωθεί επί του μοναδικού στόχου διευκόλυνση σταθερότητας και ειρήνη στον κόσμο που είναι θεμελιώδης προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής ε, πολιτικής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε ένα πρώτο γύρο από τι ομάδε που ζήτησαν το λόγο. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Υπουργό να δώσει απάντηση από πρώτο γύρο ερωτήσεων και μετά θα ακολουθήσει άλλο γύρο. Έχει κρατήσει σημειώσει, α απαντήσει στι πρώτε ερωτήσει και μετά θα ακούσει άλλου τρει συναδέλφου που θα τι θέσουν ε, τι ερωτήσει. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στην ε, όμορφη μητρική μου γλώσσα, τα βουλγαρικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας και σας ευχαριστώ που υποστηρίζετε το όραμά μας και το πρόγραμμά μας όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει αυτή η διασύνδεση με τα αναπτυξιακά προγράμματα. Αναφέρθηκε αυτό θα προσπαθήσω να ακολουθήσω στις απαντήσεις μου τη σειρά των ερωτήσεων. Πράγματι, πρέπει να σας πω ότι στο πρόγραμμά μας και στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διάφορες συγκεκριμένες πολιτικές καθώς και στην παγκόσμια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε όλα αυτά μία από τις βασικές προκλήσεις είναι να εργαστούμε για να προωθήσουμε την αντοχή των διαφορών χωρών, ούτως ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις ε, κρίσεις. Οι χώρες που είναι επιρρεπείς στις κρίσεις να μπορούν να τις αντιμετωπίζουν καλύτερα. Πιστεύει η Προεδρία ότι πρέπει να διατεθούν ειδικοί πόροι για αυτό το σκοπό. Όχι μόνο μέσω άμεσης ανθρωπιστικής βοηθείας, αλλά μέσω κατάρτισης, μέσω παιδείας, μέσω δημιουργίας θεσμών στις χώρες αυτές και μέσω της παραγωγής οικονομικής αντοχής αλλά και αντοχής με την έννοια της δυνατότητας να ανταποκρίνονται οι χώρες στα προβλήματα. Να υπάρχουν θεσμοί που θα μπορούν να αντιδρούν και να χορηγούν βοήθεια και να φροντίζουν τους πολίτες. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας, αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που θέλουμε να οδηγήσει σε καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των μέσων που διαθέτουμε, αλλά και στη βελτίωση και αύξηση της ανθεκτικότητας αυτών των χωρών. Έτσι έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα της κυρίας Ντενάνο. Ε, τα αναπτυξιακά προγράμματα είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να χρησιμεύσουν ούτω ώστε να δημιουργούνται δυνατότητες, πιθανότητες, προοπτικές και να παράγουν ένα συνέστημα ασφαλείας στις χώρες που είναι οι πηγές μετανάστευσης αλλά είναι και οι χώρες διέλευσης των μεταναστών στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και σε άλλα βήματα συζητήσεων όποτε συζητούνται τα προβλήματα ασφαλείας για την Ευρώπη και για τον κόσμο το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι συζητήσεις είναι ότι η μεταναστευτική πολιτική και η ασφάλεια και η σταθερότητα ε, είναι αλληλένδετα. Χρειάζεται εξωτερική πολιτική που παράγει ασφάλεια και τα προβλήματα παράγονται σε όλο και περισσότερες περιοχές του κόσμου. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, πώς θα πλήξουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό μέσω ανάπτυξης, παιδείας, μέσω της δημιουργίας ε, θεσμών που λειτουργούν για την ασφάλεια αυτών των χωρών και οι θεσμοί αυτοί που είναι λειτουργικοί ακούγονται σαν ε, κοινοτοπία αλλά ε, το θέμα είναι πρέπει να δώσουμε μια όθηση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορούν να θέλουμε οι ευρωπαϊκές επενδύσεις να επενδύσουν σε αυτές τις χώρες. Αν δεν αισθάνονται επιχειρήσεις ότι υπάρχει ασφάλεια σε μια χώρα και δεν έχουν διαβεβαιώσεις ότι επικρατεί το κράτος δικαίου στη χώρα, δεν θα κάνουν επενδύσεις. Τώρα στη σχέση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης, για μια ακόμη φορά να αναφερθώ σε αυτό. Μια άλλη προτεραιότητα που τόνισα κατά τη διάρκεια του γεύματος ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια και ε, η μετανάστευση. Αυτή η σχέση. Όσον αφορά λοιπόν ε, τις ερωτήσεις του κυρίου Μπορέρο Σαλμών, ε, άκουσα πολλά για τη δραστηριότητά σας. Έχετε μεγάλη εμπειρία, μπορούμε να μάθουμε από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που μας στείλατε, τις ιδέες σας, οι οποίες θα είναι πολύ χρήσιμες, οι οποίες θα συμπληρώσουν τις δικές μας ιδέες που θα εφαρμόσουμε στην ε, Προεδρία μας. Αναφερθήκατε σε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω με τα οικονομικά ζητήματα. Ανεξάρτητα από τυχόν λαμπρές ιδέες που θα μπορούμε να έχουμε, όσον αφορά τα κενά τα χρηματοδοτικά που είναι 25 δις ευρώ όπως αναφέραμε προηγουμένως αν δεν έχουμε τη σωστή λοιπόν χρηματοδότηση δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας για παγκόσμια ειρήνη, να μην υπάρχουν πόλεμοι ούτε θάνατοι από τους πολέμους προς το τέλος της Προεδρίας μας αργότερα θα γίνει το Φεβράριο ένα άτυπο Συμβούλιο για την Ανάπτυξη και θα συζητήσουμε τις ιδέες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές θα αφορούν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάπτυξη. Σας διαβεβαιώνω ότι η Προεδρία θα λάβει υπόψη της όλες τις απόψεις από αυτών των θεμάτων. Βασικός στόχος θα είναι να διευκολύνουμε την χρήση αυτών των μέσων Θέλουμε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, να έχουμε καλύτερη σχέση ε, κόστους-οφέλους και να καλύπτουμε ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων. Θα σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη των συζητήσεων και μάλιστα αφού θα έχουμε στα χέρια μας το έγγραφο το σχετικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι διότι πόροι για την παιδεία αυξάνονται κάθε χρόνο και αυτό με τη βοήθειά σας. Λοιπόν, αυτό πράγματι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα διότι ε, ένα βασικό πρόβλημα της ε, μεταναστευτικής κρίσης είναι τα κενά στην παιδεία και δεν αφορά μόνο τους, μέτα τους ε, αλλά αφορά και εκείνους που φτάνουν στις χώρες μας ως, ως πρόσφυγες το πρόβλημα της παιδείας όχι μόνο στους καταβλισμούς των προσφύγων όσον αφορά την αγροοικολογία και την έκθεση όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια έκθεση που αναμένεται να εκδοθεί το καλοκαίρι πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να φιλομετρούμε αυτές τις εκθέσεις και να τις διαβάζουμε απλώς, αλλά να μαθαίνουμε από αυτές τις εκθέσεις. Διότι πρέπει mm. να μάθουμε από τα προβλήματά μας, από τις ελλείψεις μας, ακόμα και η, ο καλύτερος δωρητής ανθρωπιστικής βοήθειας, η Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, τότε θα αποτύχει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην γίνεται μια απλή ανάγνωση των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά να τις εστερνίζονται οι διάφοροι φορείς. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα τα αγροπεριβαλλοντικά, είναι κάτι που με ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χώρα που δεν χρειαζόμαστε αναπτυξιακή βοήθεια. Είμαστε δωρητές. Αλλά ε, έχουμε διπλασιάσει τις εκτάσεις ε, και είναι που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και είναι ενθαρρυντικό. Τα προβλήματα ελλείψεως ε, τροφίμων, κακής διατροφής κλπ πρέπει να αντιμετωπιστούν και το θέμα του πολύτιμου αγαθού, του νερού πρέπει να συζητηθεί. Είναι πολύ σημαντικό το νερό για να καλλιεργούνται και τα τρόφιμα που θα θρέψουν τον πληθυσμό. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Αν λησμόνησα κάτι, σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε. Μπορώ να σας δώσω απαντήσεις αργότερα ή να σας στείλω γραπτό τις απαντήσεις αν τυχόν κάποιες ερωτήσεις δεν τις ε, κάλυψα. Ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στους επόμενους τρεις ομιλητές. Άννα Θαμπόρστκα από το ΕΛΚ. Παρακαλώ Άννα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Λίντα. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς ε, να σας ε, συγχαρώ και να σας ευχηθώ για την πρώτη σας Προεδρία και παράλληλα να σας ζητήσω και συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή της παρουσίασής σας εδώ. Η ερώτησή μου. Είναι η εξής. Από πέρυσι παρακολουθούμε ε, τις ήτες ε, του Ισλαμικού κράτους σε διάφορες περιοχές ε, της Συρίας και του Ιράκ. Απελευθερώθηκε η, η, το Χαλέπι, η Μοσούλη και το βαθύπεδο του, της Νινεβή. Μετά την απελευθέρωση των περιοχών αυτών βλέπουμε ότι η κατάσταση που άφησε το Ισλαμικό κράτος είναι καταστροφική. Δεν υπάρχει καμία υποδομή, δεν υπάρχει στέγαση, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό, δεν υπάρχει ηλεκτρισμός. Σχολεία, παιδεία, υγεία, τίποτα. Και φυσικά ο πληθυσμός που ε, απομακρύνθηκε από αυτές τις περιοχές για να επιβιώσει θα ήθελε να επιστρέψει. Εμείς ως Ένωση κάνουμε διάφορες συλλογές ε, πόρων. Και πολλές εκστρατείες γίνονται από μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την ανοικοδόμηση των περιοχών αυτών. Οπότε η ερώτησή μου είναι σε τι βαθμό η Βουλγαρική Προεδρία προβλέπει πρωτοβουλίες για να βοηθήσει οικονομικά τις περιοχές αυτές ούτως ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοί τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Και να προσθέσω. Και αυτό που συμβαίνει στο Ίντλιπ τώρα, κοντά στα τουρκικά σύνορα. Πολλοί από τις περιοχές που αναφέρατε πήγαν τώρα εδώ. Και τώρα ε, πρέπει να ξαναφύγουν γιατί η σύγκρουση έχει φτάσει σε αυτή την περιοχή της Συρίας. Μπορούμε λοιπόν να αναμένουμε μία ακόμη ανθρωπιστική κρίση. Καλύτερα λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι. παρά να αντιμετωπίζουμε τελευταία στιγμή την κατάσταση. Νόρμπερτ Νόιζαρ. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις απόψεις μας μαζί σας. Λοιπόν, μερικές παρατηρήσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο συνάδελφος Ενρίκε, που είναι και παΐων, είπε πολλά, αλλά είπατε σαφώς ότι το, ανθρωπιστικό, το χρηματοδοτικό κενό για την επίλυση των ε, κρίσεων μεγαλώνει και αυτό επειδή η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς έχει κάνει περικοπές. Και απαιτεί επίσης ε, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τον, ε, τη συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό του οργανισμού αυτού. Υπάρχει λοιπόν μία αντίφαση. Μία τόσο πλούσια χώρα όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε μειώνει την ε, συμμετοχή της στην αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων, παράδειγμα Παλαιστίνη, ενώ ζητεί από όλους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Για τον τομέα της εκπαίδευσης, βεβαίως σωστή προσέγγιση αυτή, πρέπει κυρίως να εστιάσουμε ιδιαίτερα στους καταβλισμούς ε, προσφύγων, να μην χάνουν τα παιδιά την εκπαίδευσή τους. Γιατί θα χάσουμε μια ολόκληρη γενιά. Θα μείνει αμόρφωτη και η, η μόρφωση παίζει μεγάλο ρόλο. Ιδίω για ε, πρόσφυγες, οι οποίοι αν δουν τα παιδιά τους δεν έχουν καμία προοπτική. Εάν δουν δεν έχουν καμία προοπτική θα έρθουν και αυτοί στην Ευρώπη. Επίσης για την εφαρμογή των ε, βιώσιμων ε, στόχων για την ανάπτυξη. Αυτό δεν ε, απευθύνεται μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στα κράτη-μέλη. Θα έπρεπε σχετικά σύντομα να περάσουμε στη φάση εφαρμογής των στόχων αυτών. Και συγκεκριμένα κάθε κράτος μέλος να δεσμευθεί. Κατά την Προεδρία σας θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση για την συμφωνία του Κοτονού μετά το 2020 και χαίρομαι που θα φιλοξενήσετε την ε, ισομερή συνέλευση ΑΚΕΟΚ γιατί πολλά κράτη-μέλη κατά την Προεδρία τους ε, αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν αυτή τη διοργάνωση και είπαν να γίνουν στι Βρυξέλλες. Είναι πολύ πιο θετικό να εμπλέκονται περισσότερο τα κράτη-μέλη. Πέρυσι χαίρομαι που ε, και η Μάλτα φιλοξένησε αυτή τη διοργάνωση και χαίρομαι που θα συνεχίσετε αυτή την παράδοση που ξεκίνησε η Μάλτα. Και κάτι για την ε, μεταναστευτική πολιτική. Η Βουλγαρία βεβαίω έχει μακρά εξωτερικά σύνορα. Και υπάρχει εδώ έλλειψη αλληλεγγύης έναντι της υπόλοιπη Ευρώπης γιατί δεν γίνεται σωστός έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα. Και ίσως η σημερινή κατάσταση να επιδεινώσει το πρόβλημα. Γιατί ξέρετε πως είναι η κατάσταση και στα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να επιδεικνύουν αλληλεγγύη. Και εμεί πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη με τη Βουλγαρία βεβαίω. Γιατί η Βουλγαρία βεβαίω ε, γενναιόδωρα υποδέχεται τα άτομα που διώκονται. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που μόλι έμαθα. Η χώρα σα για 75 χρόνια κάτω από πολύ δύσκολε καταστάσει, πριν από 75 χρόνια, με συγχωρείτε, και συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 43 αρνήθηκε να ε, αποσταλούν από την χώρα στα στρατόπεδα εξολόθρευσης ε, οι Εβραίοι. Τους προστατεύσατε. Αυτή σας η παράδοση νομίζω σας εμπνέει και τώρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης των προσφύγων. Ευχαριστώ πολύ. Η Σεσίλ Κέγκε. Ευχαριστώ Λίντα. Ευχαριστούμε και εσάς κύριε Υπουργέ. Πρώτα πρώτα. Θα, θα ήθελα να εκφράσω την ελεγγύη μου προς ε, ε αυτούς τους ακτιβιστές του Save the Children που υπέτσαν αυτή την επίθεση μέσα στην αποστολή τους. Εκεί που βοηθούν τα παιδιά. Αυτή είναι η αποστολή τους και ακριβώς γι' αυτό τους επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν και οπότε έχουν την αλληλεγγύη μου. Και είναι τόσοι πολλοί οι θελοντές. όλοι αυτοί που συνεργαστούν, συνεργάζονται και ζουν μέσα σε ανασφάλεια. Ε, πολλές φορές απαράγονται, δεν έχουν καμία προστασία. Ε, γι' αυτό και με ε, αυτές τις ε, συνθήκες που εργάζονται και δεν είναι μόνο στο Αφγανιστάν το Save the Children, είναι τόσοι πολλοί. Πρόκειται για ε, μεγάλη προσπάθεια που έχει πέσει σε αυτό τον τομέα. Θα πρέπει να σκεφτούμε αυτούς που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην βοήθεια των άλλων. Είναι 250 εκατομμύρια ε, αυτοί που έχουν ε, ανάγκη και πάρα πολλοί από αυτούς είναι παιδιά. Και τι είναι ο μετανάστης, κάποιος που θέλει να έχει μια καλύτερη ζωή, είναι κάποιος που αναζητάει καλύτερο μέλλον. Οπότε όντως θα πρέπει να συνδεθεί η ανθρωπιστική βοήθεια με την ανάπτυξη. Αλλά να μην χρησιμοποιούμε αυτή, αυτό τον συσχετισμό χωρίς να έχουμε κάποιο είδους μακρόπνο σχεδιασμό. Χρειάζεται αυτή η πολιτική της ανθεκτικότητας πολιτικά, οικονομικά, για το κλίμα. Άρα εκεί θα πρέπει να κατατείνουν προσπάθειές μας. Αυτό το θέμα είναι ένα ανοιχτό κεφάλαιο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς από εκεί ξεκινάει η ανάπτυξη και η κυριαρχία κάποιας χώρας. Πρέπει όμως να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες που μέσα, σε έναν, ε, μέσα από έναν πόλεμο ε, που έχουν βγει από αυτόν και τώρα έχουν κάποια κρίση. Άρα με αυτή την πολιτική της ανθεκτικότητας να βοηθήσουμε. Έτσι μόνο αυτές οι χώρες θα μπουν στην ανάπτυξη. Άλλο τρίτο θέμα. Οι εμπόλεμες ζώνες είναι πάρα πολλές. Λέμε για την Ιεμένη, ε, το Κονγκό, την ε, Σομαλία. Σε τόσες χώρες έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ε, λοιμός. Και μην νομίζουμε ότι αυτό είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν μην το ξεχνούμε. Και έχουμε πει και αυτέ τι ε, λεγόμενες κρίσεις χαμηλή έντασης. Ε, δεν μου αρέσει να εγκαταλείψουμε ε, αυτό τον ε, όρο. γιατί απλώς πρόκειται περί πολέμων όπου σκοτώνονται άνθρωποι και είναι τόσε χώρες όπου έχει καταστεί κάτι το χρόνιο ο πόλεμος η η κρίση. Άρα θα πρέπει με ένα ταμείο να βοηθήσουμε αυτούς που τόσο δυσκολεύονται που χάσαν το σπίτι τους που δεν μπορούν να γυρίσουν στον τόπο τους. Και τώρα κάτι τελευταίο όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια κάτι το οποίο για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε στην ε, Ευρώπη ε, και στην Ιδωμένη, στον Βαλκανικό Δίωπης Βαλκανική Διαδρομή. Ανθρωπιστική κρίση μέσα στην Ευρώπη. Ε, σίγουρα αυτόν λάβουμε υπόψη για τη σημερινή προσέγγιση στο θέμα αυτών που ζητούν άσυλο. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Νόρμπερτ. Και ε, επίσης στο ότι έχουμε από Αφρική, Καραβική και Ειρηνικό όσους συμμετέχουν στην Ισομερή Συνέλευση ΑΚΕ από εκεί μπορεί να βγει μια εταιρική σχέση που όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρος. Δεν έχει ζητήσει άλλο τον λόγο. Τους Παλαιστίνους δεν είπαμε τίποτα και είπαμε ότι έχουμε θέσει σε 90 χώρες από Ευρώπη και Ασία που στρέφονται τώρα προς την Παλαιστίνη που ξέρουμε τι γίνεται εκεί με τους πρόσφυγες. Είχα πάει στην Δυτική Όχθη τον Νοέμβριο. Και ιδίω όσα γίνονται στην Γκάζα είναι τρομερά, φοβίζουν. Και ξέρετε, το κατά κεφάλι εισόδημα είναι 3.000 δολάρια και χίλια στην Γάζα όπως και στο Κονγκό. Και πολύ λίγοι τρέχουν την άδεια να πάνε να βοηθήσουν τους τραυματίες. Υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Πολλές φορές 22 ώρες την ημέρα δεν υπάρχει νερό στη Γάζα. Ε, κανένα δεν συμφέρει να συνεχιστεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Έχει κάποιο πρόγραμμα σχετικό ο ΟΗΕ, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Τι είναι αυτό, είναι κάτι σαν, να μας κούρασε το Παλαιστινιακό, μα δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Ούτε το Συμβούλιο έχει τη σχετική συζήτηση. Άρα θα πρέπει να στραφούμε στο πρόβλημα αυτό. Να μην γίνει ανθρωπιστική κρίση, πολιτική κρίση. Αρκετές έχουμε στον κόσμο. Χειροτεύουμε όλα τα πράγματα. Οπότε το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Πολύ σημαντικό. Όχι, ούτε στην Επιτροπή μας. Το έχουμε συζητήσει όσο θα έπρεπε. Ελπίζω να το προσέξει το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ζαχαρίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση. Το συζητήσαμε αυτά τα θέματα τη Δευτέρα. Και στο γεύμα που το συζητήσαμε αυτό και διαβεβαιώσαμε ότι τον πρέσβη της Παλαιστίνης ότι θα αυξήσουμε τη βοήθεια προς τη Γάζα. 6 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ε, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι, τα συζητήσαμε αυτά τη Δευτέρα. Και θα αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το λαό της Γάζας. Αυτό το συζητήσαμε και με την στα πλαίσια της Διακοινοβουλευτικής ε, Επιτροπής για την Παλαιστινιακή Συμφιλίωση είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εκτός μικροφώνου η πρόεδρος. Συγγνώμη κύριε Υπουργό. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι δεν μπόρεσα να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων, αλλά κάποιες από αυτές ανήκανε στο μεγάλο, στο γενικό παζάρι, όπως αποκαλείται, δεν είναι σωστός ορισμός αυτός, αλλά παρόλα αυτά ε, το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που επιτεύχθη το 2016 στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, στην οποία συμμετείχαν 3.600 συμμε... Ε, συμμετέχοντες, αν εφαρμοστούν τα συμπεφωνημένα, τότε αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση της αποδοτικότητας και θα δημιουργούσαμε νέες μεθόδους καινοτόμε για να χρησιμοποιούνται όλοι οι πόροι συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα για να καλύπτεται η ζήτηση. Ας είμαστε ειλικρινεί. Αρχίζουν και σωρεύονται οι κρίσεις. Κάποιες είναι ανθρωπογενείς, κάποιες είναι αποτελέσματα φυσικών καταστροφών. ανεξάρτητα από την αύξηση της βοήθειας από τον ιδιωτικό ή τον κρατικό τομέα. Πιστεύουν πραγματικά ότι αν δεν έχουμε αποτελεσματικότερο σύστημα μέσω των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων του φορέα που χορηγεί τη βοήθεια χρησιμοποιώντας επιστημονικά επιτεύγματα, νέα τεχνολογία, καινοτομίε για να πετυχαίνουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας τίθενται. Διαβάζοντας την έκθεση του 2017 των Ηνωμένων Εθνών που αφορά την υλοποίηση του σχεδίου δράσεως που απέρευσε από τη Σύνοδο Κορυφής Κωνσταντινούπολης ε, του 2016, τη Μεγάλη Συμφωνία, παρόλο που είμαστε στην πρώτη γραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε καλύτεροι όσον αφορά το να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, δεν πρέπει να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι παρόλα αυτά. Αντιθέτω, πρέπει την ορμή που δημιουργήθηκε να τη συντηρήσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και αυτά που κάνουμε τώρα δεν αρκούν. Όταν μιλάμε για λησμονημένες κρίσεις, ναι, η Βουλγαρική Προεδρία έχει κάποιες ιδέες για την αντιμετώπιση τους. Κάποιες από αυτές αναφέρθηκαν από εσά εδώ στην αίθουσα. Εγώ θα έλεγα ότι η Συρία είναι μια περιοχή όπου σοβεί κρίση επί μακρών. Και δεν είναι ελκυστική πια για τα ΜΜΕ και οι μόνοι που συνεχίζουν να αναφέρουν το πρόβλημα είναι αυτοί που συζητούν με αυτή την Επιτροπή ε, ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική. Στο ευρύτερο, για το ευρύτερο κοινό ε, είναι μια κρίση η οποία είναι συνηθισμένη και γι' αυτό δεν υπάρχει απαραίτητη κατανόηση για τα προβλήματα στην κοινωνία. Λοιπόν, το Ιράκ, άλλο ένα παράδειγμα, η Εμένη, η Λιβύη, λησμονημένες κρίσεις, Νότιο Σουδάν, το Κονγκό, η Δημοκρατία του Κονγκό, Αυτές είναι χώρες που έχει εντοπίσει η Βουλγαρική Προεδρία, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν αυτές τις συζητήσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο συγκεκριμένο φόρουμ που θα λάβει η χώρα. Σχετικά με την παιδεία, που συνεχώς αναφέρεται σαν θέμα, είναι αποδεδειγμένο ότι ένας από τους βασικούς στόχους της γενικότερης στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ένας από τους στόχους της χιλιετίας είναι να εξασφαλίσουμε το ότι μέχρι το 2030 κάθε παιδί που θα γεννιέται οπουδήποτε στον κόσμο θα έχει πρόσβαση σε ποιοτική παιδεία. Εγώ δεν μπορώ να θέσω την προτεραιότητα των στόχων, αλλά πιστεύω ότι αυτή η παιδεία είναι προαπαιτούμενο για να εφαρμόσουμε και να πετύχουμε τους άλλους στόχους της ε, χιλιετίας. Όσον αφορά λοιπόν την υλοποίηση των διαφόρων μέτρων σε κάθε χώρα, λυπούμε, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ εκτενώς στις διάφορες λεπτομέρειες. Εμείς σαν ε, Προεδρία ε, δεν μπορούμε να πούμε σε κάθε κράτος μέλος πού να εστιάσει την προσοχή του, σε ποιο στόχο. Γενικά χρειάζεται πιο συντονισμένη προσέγγιση. Πρέπει να συνεργαστούμε τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τα κράτη-μέλη και με, τους, με τις διάφορες υπηρεσίες τις επιφορτισμένες με αναπτυξιακή ε, βοήθεια ε, και έτσι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Όσον αφορά τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε για τη Βουλγαρία ως χώρα και τους Βουλγαρούς. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι επίτευγμα του βουλγαρικού λαού, της βουλγαρικής εκκλησίας και φέτος θα γιορτάσουμε 75 χρόνια από τότε που σώσαμε τους ε, Εβραίους της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία είναι η μόνη χώρα ε, που δεν απέλασε κανέναν από τους Εβραίους ε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και αυξήθηκε ο εβραϊκός πληθυσμός αυτή την περίοδο, κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ σκοτεινής περίοδου της πρόσφατης ε, ιστορίας, της νεότερης ιστορίας μας. Όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή, είναι πολύ σημαντική αυτή η περίοδος. Έχουμε ένα σχέδιο κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου του Ιουνίου και τότε ελπίζουμε να πετύχουμε συμφωνία όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή ούτως ώστε όπως σας είπα και στο γεύμα να μπορεί να συμμετέχει το Κοινοβούλιο σε όλα τα τεκτενόμενα. Ξεκινάμε από πολύ καλά θεμέλια, από πολύ καλή βάση και έχω υπόψη μου τι έγινε στο τελευταίο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Όσον αφορά τη μετανάστευση, νομίζω ότι ήδη το κάλυψε αυτό το ζήτημα. κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου απαντήσεων που έδωσα, εν κατακλείδη. Θα ήθελα, κλείνοντας, να προβώ σε μια σύντομη σύνοψη, να παρουσιάσω συνοπτικά το θέμα. Ο στόχος που έχουμε μπροστά μας, ο κοινός μας στόχος, είναι πρωτίστως να αποφύγουμε τις κρίσεις Πράγματι, οι φυσικές καταστροφές, οι θεομηνίες δεν μπορούν να αποφευχθούν, αλλά έτσι θεωρούμε, αλλά δεν πιστεύω ότι αληθεύει. Όσον αφορά όμως την αλλαγή του κλίματος ή τη διατήρηση των φυσικών πόρων, εκεί πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό μπορούμε να ασχοληθούμε με την πρόληψη, να πετύχουμε την πρόληψη και μπορούμε να αποφύγουμε τις κρίσεις με αυτόν τον τρόπο και τον αριθμό των θυμάτων των θεομηνιών. Όταν έχουμε πολύ ε, ε, δυνατές βροχοπτώσεις ή άλλες φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές, θα πρέπει να στεστούμε στο πώς θα τα αποφύγουμε αυτά. Και χαίρομαι που αυτό θα επεξεργαστούμε εξετάζοντας την σχέση μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει να βελτιώσουμε την αθεκτικότητα των χωρών και να εστιαστούμε και επί της παιδείας. Α, κάτι που δεν κάλυψα, το ξέχασα. Το ερώτημα της κυρία Αγκέγκε, τι κάνουμε για εκείνους οι οποίοι κινδυνεύουν, διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να σώσουν τις ζωές άλλων. Τι κάνουμε για τους εθελοντές. Ε, πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλες οι υπηρεσίες που εργάζονται σε αυτό το τομέα θα πρέπει να έχουν έναν βασικό στόχο και αυτό να διαφυλάσσουν τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Ταυτόχρονα ε, από όλα τα κόμματα και από όλες τις χώρες υπήρξε να υπάρχει σαφής πολιτική αντίδραση όταν βλέπουμε σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Καμιά φορά δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτό γίνεται από μεμονωμένα, αποσπασματικά από κάποιες αρχές χωρών. Πρέπει να υπάρχει μια σαφής πολιτική αντίδραση όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξεκάθαρη. Αυτά και ευχαριστώ. Δεν ξέρω τώρα αν τα κάλυψα όλα. Κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, Εάν κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν έχουν λάβει απάντηση, αντιδρούν, κουνάνε το χέρι του, ζητάνε να πάρουν το λόγο, αλλά δεν βλέπω κανένα συνάδελφο να αντιδρά έτσι. Οπότε θεωρώ ότι απαντήθηκαν τι ερωτήσει, εκτό αν κάποιο συνάδελφο θέλει να επιμείνει, να επανέλθει σε κάποιο θέμα. Κοιτάξτε, ούτω ή άλλω είναι η έναρξη μια ε, διαδικασία. Μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε πολλέ ευκαιρίε να συνεργαστούμε. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σα Ευχαριστώ τους ε, συνεργάτες σας ε, και τους υπαλλήλους του Συμβουλίου. Ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν νέες κρίσεις. Γιατί έχουμε ήδη αρκετέ για να μα απασχολήσουν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σα βοηθήσουμε στην εργασία σα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα. Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό και νομίζω να την ευχαριστήσουμε και εκείνη και του συνεργάτε τη με το συνήθι τρόπο. Θα πρέπει να προσθέσω ότι ε, με ενημέρωσε για το γεγονό αυτό ότι υπάρχει αυτή η επέτειος της αποφυγής ε, του ολοκαυτώματος στη Βουλγαρία είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι κατάφεραν να σταματήσουν την εξολόθρευση των Εβραίων από τη Βουλγαρία τουλάχιστον. Συνάδελφοι, μια πολύ σύντομη διακοπή μέχρι τις 4. Θα παρακαλώ να είστε εδώ στις 4 για να συζητήσουμε τη συνάντηση κορυφής με την Αφρική. Ελπίζω ιδιαίτερα όσοι ήταν παρόντες να ε, είναι εδώ και στις 4 για να συζητήσουμε για την περαιτέρω στρατηγική μας.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 Okay, if people can start taking their seats again, it would be helpful. Παρακαλώ καθίστε, παρακαλώ καθίστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μήπως μπορείτε να τους πείτε σε όσους είναι έξω ότι εξαρχίζουμε και βλέπω είναι λάθος το διάλειμμα γιατί πάνε για καφέ και δεν ξανάρχονται πολύ. Λοιπόν, προχωράμε τώρα αγαπητοί συνάδελφοι. Στο 14 συμπεράσματα της ε, πέμπτης ε, συνάντησης ε, κορυφής Ένωσης Αφρικής που έλαβε χώρα στο Αμπιτζάν. Διάφοροι συνάδελφοι ήσαν εκεί από την Επιτροπή μας. Υπήρξαν μια σειρά από εκδηλώσεις, συνάντηση του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, μια αντιπροσωπή από την Επιτροπή μας όπως είπα ήταν παρούσα και είχαμε χρήσιμες επαφές με Αφρικανούς κοινοβουλευτικούς που ελπίζω να βοηθήσουν. Θα συναντηθούμε αύριο στη μία με την αντιπροσωπεία του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου. Εγώ δεν θα μπορέσω να είμαι, αλλά ελπίζω να πάνε άλλοι συνάδελφοι. Λοιπόν, τι έχω να σας αναφέρω από τους Αφρικανούς κοινοβουλευτικούς. Θέλουν πολύ περισσότερη επαφή μαζί μας. Δεν θέλουν μεγάλες επίσημες εκδηλώσεις θέλουν να μπορούν να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι για να συζητήσουν συγκεκριμένα θέματα. Χθε συναντήθηκα με βουλευτές από την Κάμπια. Τώρα που έχουμε μια νέα πιο δημοκρατική περίοδο στην Κάμπια και θέλουν να συζητήσουμε πώς συγκεκριμένα θέματα, πώς κάνουμε τον κοινωνιστικό έλεγχο, πώς εγκρίνουμε τον προπολογισμό, πολύ συγκεκριμένα. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Τώρα για τα αποτελέσματα της συνάντησης κορυφής, Έχουμε ομιλητέ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Κουν Φερμπέκε, που ασκεί χρέη ε, διευθυντή για θέματα Αφρικής στην ε, ΙΕΑΣ και έχουμε τον Ντούλς που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με την Αφρική στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ. Θα μας πούν λοιπόν τι συνέβη. Και εδώ παρόντες είναι ο κύριος Ιβ Σόμβιλ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ε, των θεμάτων ε, ΑΚΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έχετε στα εγγραφά σας και μια έκθεση από την αντιπροσωπή Αντέβε της Νάδης κορυφής και την διακήρυξη του Αμπιτζάν. Πού είναι ακριβώς ε, τα πορίσματα αυτής της συνάντησης κορυφής. Διακήρυξη του Αμπιτζάν του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου και υπήρξε και μια κοινή δήλωση των Ευρωβουλευτών και των Αφρικανών Κοινοβουλευτικών. Αυτή είναι η έκκληση του Αμπιτζάν. Διάφορα λοιπόν κείμενα που λάβατε για να θέσουν τη βάση. Δεν ξέρω ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος. Παρακαλώ, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ο κύριος Φερμπάκε. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Συζητήσαμε επανειλημμένα και πριν τη συνάντηση κορυφής και είχατε και μια πολύ καλή έκθεση της κυρίας Κιέγκε που, όχι του κυρίου Πονγκά μάλλον, που μας βοήθησε για να εκπονήσουμε το πρόγραμμα δράσης και την περαιτέρω συνεργασία μας και προετοιμάζουμε και την ε, Υπουργική Συνάντηση Ένωσης Αφρικής για την οποία θα συνεργαστούμε μαζί σας. Τώρα για την ίδια τη συνάντηση κορυφής. Η εξολόγησή μας είναι ότι συνολικά ήταν επιτυχημένη. Υπήρξαν οι συνήθεις ε, οργανωτικές δυσχέρειες, δεν έρεαν όλα αλλά επί της ουσίας τονίστηκε ο μεγάλος βαθμός αλληλεξάρτησης των δύο οχθών της Μεσογείου και ανάγκη συνεργασίας. Επίσης ε, η συμμετοχή και από τις δύο πλευρές ήταν υψηλού επίπεδου. Ευρωπαϊκό επίπεδο όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλα τα κράτη-μέλη, σχεδόν όλα, σε πολύ υψηλό επίπεδο και επίσης από αφρακανική πλευράς. Πρωτόγνωρα ε, υψηλό επίπεδου συμμετοχή. Κατά τη γνώμη μας, αυτό υπογραμμίζει ότι περνάμε σε μια πιο όρημη, πιο πολιτική, πιο ισότιμη σχέση. Αυτό είναι κάτι σχετικά νέο. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτή την διάσταση χορηγού και δικαιούχου. Θέλουμε επίσης να δεσμευθούν για την επίτευξη των στόχων πολιτικής περισσότερο οι ίδιοι Αφρικανοί. Παρουσίασαν οι Αφρικανοί την, το όραμά του, το πρόγραμμα δράση τους και για την ανάπτυξη αλλά και για την μετανάστευση. Η λιβική κρίση που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της ε, συνάντησης κορυφής απέδειξε την ανάγκη οι Αφρικανοί να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον τους. Αυτό αναφέρεται στην πολιτική διακήρυξη που δηλώσατε, όπου υπάρχουν πολύ περισσότερο αμοιβέ δεσμεύσει. Κάτι για το οποίο εργαστήκαμε σκληρά και κατά τι προπαρασκευαστικέ και κατά τη συνάντηση των ε, ανωτέρων υπαλλήλων στο Αμπιτζάν, κάτι που πρόθεσε και η κυρία Μογκερίνη όταν ολοκληρώθηκε η υπουργική διακήρυξη. Η νεότης ήταν το βασικό θέμα πριν από τη συνάντηση κορυφής κάναμε πολλές προσπάθειες να ακουστεί η φωνή της νεότητας, των νέων, σε όλες τις φάσεις διαδικασίας και στη συνάντηση κορυφής. Υπήρξε μια πολύ θερμή συνάντηση μεταξύ διαφόρων αρχηγών κρατών και εκπροσώπων των νέων. Οι νέοι είχαν δικαίωμα λόγου σε όλες τις ε, εκδηλώσεις. Δεν ήταν λοιπόν μια συνάντηση κορυφής μόνο για τους νέους, αλλά και με την παρουσία των νέων η μετανάστευση τώρα είναι μια νέα διάσταση. Όχι μόνο μια διάσταση επίγουσας ανάγκης, αλλά επίσης ε, μια προσέγγιση ότι είναι κοινή μας ευθύνη. Ξέρετε ότι αμέσως μετά υπήρξε αυτή η πολιτική δήλωση μεταξύ της Ένωσης ε, των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης για την μεταναστευτική κρίση στη Λιβύη και αυτό ξεκίνησε αμέσως μετά τη συνάντηση κορυφής και συνεχίζεται για να ενισχυθεί η εθελούσια επάνωδος από τη Λιβύη στις χώρες προέλευσης και για να υπάρξουν περισσότερες ευκαιρίες για όσους έχουν ανάγκη. Μεταξύ της ε, συνάντησης κορυφής και τέλους Δεκεμβρίου 7.000 έχουν εθελουσίως επανέλθει και ελπίζουμε άλλες 10.000 να επανέλθουν σύντομα. Οπότε θα υπερβούμε το στόχο του Αμπιτζάν που ήταν 15.000. Μάλλον θα φτάσουμε στις 17. Είναι βέβαια ένα πρώτο βήμα στη συνάντηση κορυφής. Επίσης ε, θελήσαμε να υπάρξει μια πανυπηρωτική διάσταση για το θέμα αυτό. Η Αφρική τώρα λοιπόν θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι τέρος της για το θέμα της μετανάστευσης. Άλλες βασικές πρωτοβουλίες όμως δεν ε, επέτυχαν πάντα για το μνημόνιο αλληλοκατανόησης για την ασφάλεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν καταλήξαμε. Δεν ήταν ε, έτοιμη η αφρικανική πλευρά, υπήρχαν και κάποια πολιτικά θέματα. Θα πρέπει να επανέλθουμε. Ελπίζουμε και δεσμευόμεθα ότι θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες συζήτηση για το θέμα αυτό. Ξέρετε ότι είναι βασικό θέμα για τη συνεργασία μας και θέλουμε να υπάρξει επιτυχής κατάληξη. Ανέφερα τον διυπηρωτικό διάλογο για την μετανάστευση, μεγάλη επιτυχία και επιτύχαμε πολλά για τα οικονομικά θέματα, επενδυτικά σχέδια για παράδειγμα. Θα επανέλθω. Ή μάλλον θα χρειαστεί περαιτέρω δουλειά εννοούσα. Πρέπει να συνεχιστεί λοιπόν η εργασία. Η ΝΤΕΒΚΟ έχει ένα πρόγραμμα δράση, το οποίο δεν μπορέσαμε να εγκρίνουμε στο Αμπιτζάν, δεν υπήρχε χρόνο. Έχουμε ακόμη τρει μήνε. Έχουμε κάνει την ε, προετοιμασία, συζητάμε με τα κράτη-μέλη σήμερα. Και κατόπιν θα απευθυνθούμε και στην αφρικανική πλευρά για να συμβάλλουν και εκείνοι για να ολοκληρωθεί όπως ε, προβλέπετε πριν το τέλος Φεβρουαρίου. Επίσης κάποια συνέχιση της δουλειάς, η ετήσια υπουργική συνάντηση πρέπει να γίνει φέτος. Είναι λοιπόν σαφές ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να διεξαχθεί αυτή η συνάντηση. Άρα υπάρχει ειλικρινής βούληση συνέχισης του διαλόγου. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο. Μόλις το πρότεινε η Φεντερίκα Μογκερίνη, το ενέκριναν και οι δύο πλευρές. Ο μηχανισμός παρακολούθησης της συνέχειας που δίνεται. Πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά, τις αποφάσεις δηλαδή, πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά από αυτού και να συνδεθεί με τη συζήτηση για τι θα διαδεχθεί το κοτονού. Η συμμετοχή τώρα όλων των ενδιαφερομένων φορέων στην ε, παρακολούθηση της συνέχισης θα μας απασχολήσει. Δεν είναι ικανοποιητική μετά τη συνάντηση των Βρυξελών το ετήσιο κοινό φόρουμ. Θα θέλουμε μέχρι το καλοκαίρι να συμμετάσχει περισσότερο η κοινωνία των πολιτών, οι νέοι, τα κοινοβούλια. Είναι πολύ σημαντικό για να αναπτυχθεί η εταιρική μας σχέση. Ευχαριστώ πολύ και στη διάθεσή σας. Πρόεδρος. Το τελευταίο. Το κοινό ετήσιο φόρουμ. Η συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων. Στις Βρυξέλλες είπαμε ότι θα υπάρχει ένα κοινό ετήσιο φόρουμ όπου τα δύο θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη, η κοινωνία των πολιτών και άλλοι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν δεν συμφώνησαν όλες οι αφρικανικές χώρες, ιδιαίτερα η Αίγυπτος. Πρέπει λοιπόν να επινοήσουμε κάτι διαφορετικό που να είναι ρεαλιστικό. Ευχαριστώ πολύ, καταλαβαίνω λίγο πρόεδρος. Παρακαλώ, κύριε Κούν. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω, ίσως δύο λόγια από πλευράς πολιτικής. Το συζητήσαμε πριν πάμε στο Αμπιτζάνι αφετηρία μας σαφώς ήταν το να υπάρξει περισσότερη συνειδητοποίηση στην ε, Ευρώπη ότι δηλαδή λόγω της μεταναστικής κρίσης είναι πολύ σημαντική η για την Ευρώπη είτε είναι καλά είτε κακά τα, μοντάδα μαντάτα από την υπάρχουν επιπτώσεις και είχαμε αρκετά εντατική και συναντήσεις στο Αμπιτζάν. Οπότε το ψηφιδωτό έτσι συμπληρώθηκε. Δηλαδή, ότι θεωρούν οι Αφρικανοί ότι έχουν την τύχη τους στα χέρια τους. Ότι η Αφρική, εάν λάβει τις σωστές αποφάσεις, έχει μέλλον. Έχει τους φυσικούς πόρους, έχει τους ανθρώπινους πόρους. Υπάρχουν οι δυνατότητες επομένως και αυτό το έχουν συνειδητοποιήσει. Και όλη η Αφρικανική Ένωση και το κάθε κράτος χωριστά. Είναι σημαντικό αυτό να ληφθεί υπόψη. Θέλει η Αφρική να είναι παράγον σε έναν πολυπολικό κόσμο. Δεν θέλει να είναι απλώς ο στόχος παρεμβάσεων των μεγάλων παικτών και ξέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί από μόνο του. Και η σαν της κορυφής της επομένης εβδομάδας έχει στην μέση διάταξη της μεταρρυθμίσης του Καγκάμι ούτως ώστε η Ένωση να είναι πιο αποτελεσματική και εταιρικέ σχέσεις να υπάρξουν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους παίκτες. Να, πώς αποδεικνύεται το ότι βλέπουν στα σοβαρά το ρόλο Αυτό βρισκόταν στο επίκεντρο της δυναμικής που αναπτύχθηκε στο Αμπιτζάν. Νομίζω ότι εμεί ακολουθήσαμε σωστή τακτική, αλλά ξέρετε δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα. Να, ένα πάνω περιστατικό τη συζήτηση που έγινε για το πρόγραμμα εξωτερικών επενδύσεων και ουσιαστικά είναι εργαλειοθήκη, δεν είναι πρόγραμμα ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε μόχλευση. Και το όραμα μας για την Αφρική, η συζήτηση που έγινε επίσης για το EIP ήταν συμβολική σημασία αυτού του προγράμματος του σχεδίου για την Αφρική για να δείξει ότι δεσμευόμαστε έναντι των Αφρικανών για να έχουμε εξισορροπημένη λύση να καλυφθούν τα συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα, μετανάστευση, ανάπτυξη πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας, παιδεία, υγεία και βέβαια οι Αφρικανοί έχουν το δικό τους θέμα, το δική τους η ημερήσια διάταξη στη συνάντηση. Αυτό φάνηκε. Επίσης, η δήλωση διακήρυξη του Αμπιτζάν αντικατοπτρίζει ακριβώς την συμφωνία που επιτεύχθηκε το ότι συναντήθηκαν ιδέες των μεν με τους δε. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική αυτή η δήλωση. Και οπότε γι' αυτό το λόγο και θα πρέπει να πετύχουμε όσον αφορά τη συνέχιση. Τη συνέχεια πρέπει να δοθεί. Και από πλευρά μα, από πλευρά Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία, από πλευρά τη Αφρικανική Ένωση. Και άρα πάμε για να χαράξουμε τις προτεραιότητες του προγράμματος δράσης. Τώρα, όσον αφορά το τι να κάνουμε υπήρξε μια σαφής σύγκληση σε όλες τις ομιλίες και από δικής μας πλευράς και από πλευράς των Αφρικανών όσον αφορά την νεολαία και τις επενδύσεις. Τις επενδύσεις στην νεολαία. Οπότε και σαφώς πρόκειψε ότι θα προσεχθεί πάρα πολύ επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση καινοτομία, επιστήμη. Έχουν όρεξη να προχωρήσουν και εμείς επίσης θα πρέπει περισσότερο από το παρελθόν να τους βοηθήσουμε. Αυτό είναι το συμπέρασμα για το μέλλον. Ε, επίσης αυτό αφορά και την επιχειρηματικότητα. Όχι απλώς να μιλούμε για ε, τις ε, αγορές αλλά να συζητήσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και μαζί το ευρύτερο θέμα της διακυβέρνησης της διαφθοράς της κινητοποίησης των ντόπιων πόρων της ανισότητες με αυτό είναι το θεματολόγιο που καταρτήσαμε Αυτά πρέπει να καταφέρουμε. Προς το παρόν θα βάλω τελεία. Okay. Thank you for outlining the... Ευχαριστώ που τονίσατε τα δύο ζητήματα για μας. Τρεις ομιλητές έχω στον κατάλογο. Τέσσερις. No I've got. Okay, oh, sorry. Yeah, we've got four speakers indicated. Τέσσερις έχουν ζητήσει το λόγο. Μαρία Νόησο, πρώτη. Μαρία Σαλ. Μαρία. Και μετά η Σεσίλ. Μαρία, εσύ. Εσύ πρώτη. Εσύ Μαρία. Οι Μαρίες μεταξύ τους θα τα κάνουν. Όλοι θα μιλήσουν τη σειρά. Ε, κοιτάξτε, το όνομα Μαρία είναι κάτι που αρκετά συχνά ακούγεται σαν όνομα στο Ευρωκοινοβούλιο, άρα δημιουργεί μια κάποια σύγχυση. Επίσης, εγώ είμαι πληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ανάπτυξης και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για αυτά τα ζητήματα. Τρεις βασικές ανησυχίες θα ήθελα να αναφέρω. Νομίζω ότι το περιεχόμενο της συνεδριάσεως ε, περιεγράφει πολύ καλά. Είπατε ότι πολλά έπρεπε να γίνουν και πραγματικά πολλά ζητήματα συζητήθηκαν και αυτό ήταν πολύ καλό. Αλλά υπάρχουν πολλοί τομεί που χρήζουν βελτιώσεων. Οπότε για την ώρα πρέπει να καθίσουμε, να παρατηρούμε, να περιμένουμε, να δούμε τι θα συμβεί και μετά να αξιολογήσουμε την πρόοδο. Τρει εντυπώσει αποκόμισα από αυτό το ταξίδι. Ελπίζω ότι δεν θα σας ενοχλήσει αυτό που θα πω. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι υπέροχο να πηγαίνουμε στην Αφρική και μόνο άντρες να πηγαίνουν στην ομάδα, στην αποστολή. Ε, στην Ολομέλεια είχαμε μόνο άντρες εκπροσώπου του Ευρωκοινοβουλίου και αυτό δεν νομίζω ότι είναι καλό. Θα πρέπει ε, να πηγαίνουμε ε, γυναίκες πολιτικούς στην Αφρική. Να προωθούμε αυτήν την ιδέα. Αν έχετε μόνο έξι άντρες εκεί να κάνουν παρουσιάσεις και γυναίκες μένουν πίσω, δεν είναι σωστή εικόνα που θα πρέπει να προβάλλουμε. Ανταυτού, η εικόνα, η οπτική εικόνα που δίνουμε στον κόσμο αυτόν τον τρόπο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό πολύ συχνά μένει σαν εντύπωση στον κόσμο, όχι τι υπόθηκε. Αυτή η εικόνα απομένει. Και είδα το πρόβλημα αυτό και με άλλε αποστολέ κατά το παρελθόν. Αλλά με αυτό το ταξίδι προβληματίστηκα ε, όσον αφορά την κυριαρχία των ανδρών και αισθανόμουν ε, κάπω άσχημα στην Ολομέλεια. Τι έγινε. Το, είχα, ήταν το κοινό που αν παρών. Ε, κανονικά έπρεπε να μπορεί να έχει παρουσία, εδώ αποκλείστηκε. Πρέπει να το συζητήσουμε. Όταν οι επισκέψεις μας σε μια χώρα ε, σημαίνουν ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει το κοινό και όταν έχουν ταξιδέψει άνθρωποι από όλο τον κόσμο και θέλουν ε, να συναντηθούν και να συναντήσουν και μέλη των ε, ΜΚΟ Νομίζω ότι πρέπει αυτού του είδους επαφές να τις προθούμε. Πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό όταν κάνουμε αυτού του είδους αποστολές. Να προσέξουμε λοιπόν ε, ούτως ώστε να μην χάνονται αυτές οι ευκαιρίες. Πρέπει να καθίσουμε και να δούμε τι ακριβώς ε, γίνεται ε, επί τόπου. Λοιπόν, και εγώ συμμετείχα στις διάφορες επισκέψεις και τα έργα που είδαμε ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα από τη φυτεία μπανάνας, την μπανανοφυτεία μέχρι ε, ε, αυτό που είχαν κάνει οι, οι Ευαγγελικοί, οι ιερείς. Ας πούμε βλέπαμε κάποιο σπίτι, απλό σπίτι, ε, η καλύβα κάποιου. Να πηγαίνουμε από υπέροχο παράδειγμα σε άλλο υπέροχο παράδειγμα, σχηματίζεται η εικόνα, τα πάντα λειτουργούν θαυμάσια. Όμως, εάν αντιθέτως πηγαίνεις και συναντάς πραγματικούς ανθρώπους και όχι αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αναμειγνύονται σε αυτού του είδους ε, τα υπέροχα προγράμματα, ε, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Δεν θέλω να φεύγω από μια χώρα και να μην ξέρω πώς ε, κινείται και ζει ο απλός άνθρωπος στα πραγματικά του, στα, στην καθημερινότητά του, στα σπίτια του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να συναντήσουμε τους απλούς ανθρώπους. Διότι θέλουμε να δούμε βέβαια τα θετικά παραδείγματα, θέλουμε να τα προβάλλουμε, να τα συζητήσουμε και να τα γνωστοποιήσουμε στον κόσμο αν είμαστε στην υποδειγματική ε, εκμετάλλευση, στο υποδειγματικό σχολείο όπου είναι θαυμάσια αντιμένοι, όλοι είναι πολύ ευχαριστημένοι, αλλά είναι ένα μικρό μόνο τμήμα, δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Όταν κάνουμε ταξίδια, ξέρω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να το οργανώσουμε, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε την πραγματικότητα και όχι μόνο τα υποδειγματικά προγράμματα. Εκεί πάντα μας καλούν. Δεν μπορούμε να φύγουμε από τη χώρα χωρίς να δούμε και λιγάκι την πραγματικότητα και ιδιαίτερα ακριβώς ε, σε αυτήν την αποστολή είχα την εντύπωση ότι επισκεφθήκαμε θαυμάσια προγράμματα ήταν σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε, αλλά θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να δω και λίγο πίσω, στα παρασκήνια. Αυτό που είδαμε ήταν μια σκηνοθεσία. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ Μαρία. Κάποια από τα θέματα διοργανώσεως των επισκέψεών μα πρέπει να συζητηθούν στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν θα πάσα αύριο, έχει συνεδρίαση στις μία. Ναι, ήταν θέμα αυτό. Σαλ Γκέρενς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με τα μεγίστης ε, προσοχής τους προλαλήσαντες. Δεν αμφισβητώ επουδενή την καλή βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως Αφρικής. Το προσπάθησαν πολλοί επίτροποι, κυρίως ο Λούι Μισελ. Κινήθηκε σε αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα επηρεάζει αυτή η εργασία τις σχέσεις με την Αφρική. Τι με ανησυχεί. ο πλουραλισμός που επέδειξε το Συμβούλιο. Ξέρουμε τις σκέψεις των μεν, αλλά τις υποσυνείδητες σκέψεις των αλλωνών, τις κρυφές σκέψεις των αλλωνών. Οι μεν θέλουν να προωθήσουν σε εμπορικές σχέσεις, να έχουν μια μεγάλη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ενδεχομένω μέσω ενός σχεδίου Marshall. Αυτό που μου λείπει όμως, σαν υπέρμαχος της ανάπτυξης, είναι η εξέταση των θεμάτων από την οπτική γωνία της ανάπτυξης, πώς θα μειωθούν οι ανισότητες, τι κριτηρία θα κινητοποιήσουμε για να αξιολογήσουμε με την πραγματική αξία της πραγματοποιηθήσεως πρόδους. Εάν ξεκινήσουμε τη διαδικασία αυτή και το Αμπιτζάν ήταν σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει ήδη να καθορίσουμε τις προδιαγραφές της αξιολόγησης τι θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, όσον αφορά την κατανομή του πλούτου, όσον αφορά τη βελτίωση της κυβερνήσεως, όσον αφορά τη μείωση της διαφθοράς και σχετικά με αυτό είχα καταθέσει μια πολύ σημαντική μαρτυρία. Μάλλον από την Ανατολική Νιγηρία ήρθε κάποιος από την επαρχία και μου από μια περιοχή που έχει αυτονομία και εκεί έχουν καταφέρει και έχει καταπολεμηθεί ριζικά η διαφθορά εκεί πέρα και ο κόσμος δεν φεύγει από εκεί, δεν μεταναστεύει γιατί έχει πιθανότητες, έχει δυνατότητες να παραμείνει εκεί γιατί έχει καταπολεμηθεί η διαφθορά. Πέρα από τις μεγάλες υποσχέσεις όπως το Αμπιτζάν πρέπει να δούμε όχι σε κάθε λεπτομέρεια αλλά σφαιρικά το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα και κάτι άλλο με ανησυχεί. Κάποιοι ακολουθούν χρηστική προσέγγιση. Κάποιοι που είναι σε αυτή την κατάσταση, κά, κάποιες χώρες. Για κάποιους κάνουν μια προσέγγιση για να λύσουν με τα δικά μας προβλήματα. Έχουμε κοινά συμφέροντα στον αφορά την ασφάλεια, αλλά κάποιοι έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Τώρα, η ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είχε προτείνει να είναι στο πλευρό της Αφρικής για να διεκδικήσει μια έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, ε, του ΟΗΕ. Αν πάρουμε τη σύγκρουση στη Λιβύη, τι έλειψε εκεί. Ε, κάποιος που να μιλήσει εν ονόμα της Αφρικής στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Τι περιμένουμε. Σε 30 χρόνια θα είναι 2 δισεκατομμύρια κάτοικοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η, η, η Ήπειρος, η Ρωσία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τρεις έδρες μόνιμες στο Συμβούλιο Ασφαλείας η Ευρωπαϊκή Ήπειρος η γυράσκουσα και έχετε από την άλλη πλευρά από την άλλη πλευρά της Μεσογείου μια Ήπειρο η οποία ε, περνάει μια δημογραφική έκρηξη. Και θα πρέπει ο Επίτροπος υπεύθυνο για την ασφάλεια, μάλλον η Επιτροπή που ε, ασχολείται με τα θέματα ασφαλής Αφρικής, να κινηθεί πιο υπεύθυνα και να αντιμετωπίσει το θέμα πιο υπεύθυνα της ασφάλειας. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν να σημειωθεί κάποια πρόοδος εκεί. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφερθεί στη συνύπαρξη σχέσεως Ευρωπαϊκής Ενώσεως Αφρικής από τη μια και τις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική συμφωνία του Κοτονού από την άλλη. Όταν συνομιλούμε με την Αφρική στο Αμπιτζάν θεωρούμε ότι όλη η αφρικανική πλευρά, όλες οι αφρικανικές χώρες ανήκουν εκεί και αυτές της Βορείου Αφρικής. Και νομίζω ότι αυτό ακολουθεί κάποια λογική. Το πρόβλημα της ασφαλείας είναι το πρόβλημα κατά της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών. Δεν μπορούμε όμως να εξαιρέσουμε το Μαρόκο, τον Ήγυρα, τον Μαλί, την Μπουρκίνα Φάσο, την Τινησία, την Αλγερία θα πρέπει αυτή την περιοχή να τη δούμε συνολικά. Αν ασχολούμεθα με το πρόβλημα στο σύνολό του σε ένα πλαίσιο και κατακαιρματισμένα σε άλλο πλαίσιο, αυτό δεν έχει νόημα. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε κάποια τάξη, να υπάρχει κάποια συνοχή. Η προηγούμενη ομιλήτρια μας είπε ότι μας δείχνουν τα έργα που είναι η δόξα της συνεργασίας μας. Μπορούμε να το γενικεύσουμε αυτό. Αυτού που συν, ε, συνήθως επισκέφτονται την Αφρική έχουν αρνητική ε, εικόνα. Πολλά έργα λειτουργούν καλά, αλλά πολλά πράγματα δεν λειτουργούν καλά. Και πρέπει να αναπτύξουμε στρατηγικές όσον αφορά την ασφάλεια. Πέρα από τα δικά μας συμφέροντα πρέπει να κοιτάξουμε. Συζητήσαμε τον Μπουρούντι, την ασφάλεια στην περιοχή των μεγάλων λιμνών, την έλλειψη κρατικών θεσμών στα βάθη της ε, δημοκρατίας του Κογκό. Τι κάνουμε με όλα αυτά τα παραπέοντα κράτη όπου δεν πρέπει, δεν λαμβάνεται υπόψη ο πολίτης. Δεν μπορούμε να κυβερνούμε τις χώρες αυτές αντικαθιστώντας τις κυβερνήσεις. Τι γέφυρες μπορούμε να χτίσουμε ούτω ώστε οι κυβερνήσεις να είναι πιο υπεύθυνε, να εθετήσουν πιο υπεύθυνε πολιτικές. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που έχω. Σχόλια. Να και να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής ε, Ενώσεως που έκαναν μισαγωγή στο θέμα. Η Βαρία Χόιμποκ και μετά η Σεσίλ και μετά θα ακούσουμε εκπρόσωπο τη ε, οικονομική συνολική Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Να ασχοληθώ με το τελικό κείμενο. Από ό,τι μάθαμε καθυστέρησε η έκδοσή του. Ήταν μόνο θέμα καθυστέρησης. Κάτι έγινε και αργήσανε ή μήπω υπήρξαν ε, διαφορετικές προσεγγίσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν και αν όντω ισχύει κάτι τέτοιο θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα ποιε διαφορές απόψεων υπήρξαν για ποια σημεία χρειάστηκαν περαιτέρω συζητήσεις και πού χρειάστηκε να αποχωρήσουν οι μεν και οι δε για να επιτευχθεί συμβιβασμό. Η Αφρικανική Ένωση δηλαδή, και οι Αφρικανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αφρικανοί. Θα ήθελα πραγματικά να μάθω για αυτά γιατί επισήμως δεν τα μαθαίνει βέβαια κανείς αυτά. Επίσης, ο Επίτροπος Νίμιτσα έστειλε ένα Twitter από τα Αμπιτζάν για την σχέση μας μετά το Κοτονού ε, αυτό με εκπλήσει γιατί η Αφρικανική Ένωση δεν έχει εκφραστεί από αυτού. Δεν ξέρω θα υπάρξει κάποια επίσημη ε, άποψη μετά την συνάντηση που θα γίνει τέλη του τρέχοντος μήνα. Τώρα, από ό,τι είδα στη διαπραγματευτική μας θέση για τη συζητήση για μετά το Κοτονού, λένε ότι οι διάφορες πυλώνες της Αφρικής θα αντικαταστήσουν τη συνολική αντιμετώπιση που υπάρχει μέχρι τώρα. Σε αυτή την ε, πρόταση καταλήξαμε από κοινού με τους Αφρικανούς, την Αφρικανική Ένωση, γιατί έχουμε μιλήσει πολύ για μια εταιρική σχέση. Αυτή είναι κοινή θέση ή αυτή είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι ακόμη. Το ανέφερε και η Μαρία Νόχλατς. Και εμείς ε, ως πράσινοι λυπούμεθα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η κοινωνία των πολιτών. Δεν τους επιτράπει να συμμετάσχουν στην πραγματική συνάντηση κορυφής. Είναι αντίθεση αυτό εφόσον θέλουμε να υπάρξει εταιρική σχέση μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ένα ένα δείγμα ότι οι δυνατότητες συμμετοχής ε, της κοινωνίας των πολιτών περιορίζεται. Αυτό το παρατηρήσαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι δυνατόν να ε, το επιτρέψουμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και η υπηρεσία εξωτερικής δράσης και οι κομισιόν το καταλαβαίνουν αυτό και θα λάβουν μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό. Συζητήσατε για τη συνάντηση των εμπλεκομένων ε, φορέων εδώ στις Βρυξέλλες που δεν διεξήχθη όπως είχε προβλεφθεί. Δεν είναι δυνατόν εμείς απλώς να κάνουμε μια συνάντηση των ενδιαφερομένων φορέων όταν γίνεται κάπου αλλού στον κόσμο η πραγματική συνάντηση της κορυφής. Πρέπει εκεί να υπάρχουν πλατφόρμες για την έκφραση της κοινωνίας των πολιτών. Διότι η ανάπτυξη και των πιο φτωχών ε, χωρών αλλά και συνολικά της Αφρικής μπορεί να συμβεί μόνο αν συμμετάσχουν οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών. Δεν θα συμμετάσχουν μόνο κάποιοι κοινοβουλευτικοί ή κάποιε επιτροπέ και δεν ξέρω εγώ τι. Χρειαζόμαστε του πολίτε που ζουν στι χώρε αυτέ. Άρα θα πρέπει να του επιτρέπεται συμμετοχή σε αυτέ τι συναντήσει. Και πρέπει να έχουν δυνατότητα να εκφραστούν. Να υπάρχει κάποια πλατφόρμα για να εκφραστούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μαρία. Η Σεσίλ Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τους δύο εισηγητές για την ενημέρωση που μας έκαναν. Είναι θετικό το ότι μπορούμε σε τακτήρια διαστήματα να τα λέμε, να ενημερωνόμαστε όπως τώρα για το Αμπιτζάν. Θα πρέπει όμως να τα πούμε πιο συγκεκριμένα. Αφετηρία έχω αυτό το οποίο είδαμε επί το... και συμφωνώ με την συνάδελφο τη Μαρία που είπε ότι θα πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα επί τόπου στις αποστολές. Να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέραν των ε, οργανωμένων προγραμμάτων και έργων. Τι γίνεται με τον κόσμο να πάμε στην πιο μεγάλη λαϊκή συνοικία του Αμπιτζάν. Να δούμε τι κάνουν οι νέοι, τι project έχουν. Εκεί που μένουν στο σπίτι τους. Να δούμε τι έχουν πετύχει με αυτά τα έργα. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν επιστρέψει από την Λιβύη που διηγούνται τις εμπειρίες τους. Είναι αυτοί που ε, θέλουν να τους ακούσει, να τους αφουγκραστεί η κυβέρνηση. Εκεί που σε κάποιο σημείο μέσα από την πόλη περνάει ένας αυτοκινητόδρομος. Δεν έχουν που να πάνε αυτοί οι νέοι άνθρωποι. Και μας είπανε αυτοί ότι έχουν μπροστά τους αδιέξοδο έτσι. Οπότε αφού θεωρούν δεν έχουν μέλλον εκεί, έτσι παίρνουν το δρόμο της μετανάστευσης και πάνε στην Λιβύη. Άρα αυτό θα πρέπει να δούμε. Τι γίνεται με την Task Force, τι γίνεται με την Εκένωση. Δεν είναι δυνατόν να εκτοπίζονται αυτοί οι άνθρωποι να πρέπει να φύγουν από εκεί που μένουν χωρίς εναλλακτική. Όντως να τους πάρουμε από την Λιβύη αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει να μπορούμε επομένως να έχουμε μια παρέμβαση εκεί επί τόπου στην πατρίδα τους. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει και για την ανεξαρτησία χειραφέτηση των γυναικών. Πήγαμε γι' αυτό το λόγο λοιπόν σε κάποια άλλη φτωχή περιοχή. Εκεί είδαμε τι γίνεται με αυτό το Ταμείο Εγγύησης για την χειραφέτηση των γυναικών είναι ένα σύστημα χρηματοδότησής τους. Πολλές φορές το αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, αλλά όμως και με αυτό το σύστημα καταφέραμε τους δώσουμε την εξαρτησία, καταφέρανε να έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις, φτιάξαν ένα σύστημα που είναι ανεπίσημο και λειτουργεί. Για αυτά τα μικρά έργα που υποστηρίζονται οι γυναίκες, κάποιοι που έχουν περιθωριοποιηθεί από το υπάρχον κατεστημένο σύστημα. Να δούμε τι γίνεται και με τις εξωτερικές επενδύσεις. Να δούμε πώς θα αλλάξουν οι λεπτομέρειες που διέπουν αυτές τις επενδύσεις. Αλλά όμως αυτά τα πρόσωπα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους. Πολλές φορές δεν ξέρουν ότι υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Και μιλήσαμε με αυτούς που ήρθαν από τη Γκάμπια. Να τους πούμε με τι μηχανισμούς μπορούν να έχουν κάποιο είδου διορθωτικέ μεταρρυθμίσεις σε οικονομία, πολιτική, ε, για τη δημοκρατία. Δεν ξέραν τίποτα. Ήταν στο σκοτάδι. Οπότε έτσι να τους ε, μαζέψουμε, να ανταλλάξουμε πληροφορίες και να μην έχουμε κάποια γραφειοκρατία. Να είναι ανοιχτό αυτό το σύστημα, αυτή η πρωτοβουλία. Έτσι θα αποκτήσει αυτή την ανθεκτικότητα η περιοχή. Α, άλλα δύο θέματα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για την διασπορά δεν άκουσα τίποτα να λέτε σχετικά με αυτό. Και είπαμε στις διακοινωνικές επαφές ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα. Τώρα τι γίνεται στο διάστημα μετά την Κοτονού και μιλήσαμε επομένως και με τους χειροβητικούς από άλλες ε, χώρες και είπαμε ότι θέλουν κάποιες ε, ισχυρές δομές θεσμικές για να μπορούν να αποκτήσουν θεσμούς στεγανούς στη χώρα τους. Δεν ισχύει σήμερα. Πόσο μάλλον όσον αφορά τα κοινοβουλιά τους. Um, Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Σομβίλ. Κύριε Σομβίλ, είστε ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής. Είπαμε ότι πέραν αυτή της συνάντησης κορυμή παράλληλα έγινε αυτή η συνάντηση των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων. Για αυτά θα μας μιλήσετε. Έχετε την σκητάλη κύριε Σομβίλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε για να σας πω ποια είναι τα αποτελέσματα των συναντήσεών μας των οικονομικών και κοινωνικών φορέων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Αφρικανικής ε, Ένωσης. Μέσα Νοεμβρίου έγινε, 15 μέρες πριν τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως Αφρικής στο Αμπιτζάν. Οργανώνουμε αυτού του είδους τις συνεδριάσεις από το 2014, αλλά είναι η πρώτη φορά όπου διοργανώσαμε αυτή τη συνεδρίασή μας πραγματικά με ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο σε αυτή την περίπτωση με το Οικονομικό Κοινωνικό Συμβούλιο περιβαλλοντικό ε, και πολιτιστικό της ακτής του Ελεφαντοστού. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία για αυτό το θεσμό ε, να προβληθεί σε αυτή την εκδήλωση. Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως είχαμε κοσόπου της ΕΚΟΣΟΚ ε, της Αφρικανικής Ένωσης αλλά των οικονομικών και κοινωνικών συμβουλίων όλων των χωρών της Αφρικής ήταν πολύ καλή συζήτηση μεταξύ στελεξικών, συγκαλιστών, γεωργών, εκπροσώπων διαφόρων επαγγελμάτων κλπ. Συνοπτικά να παρουσιάσω τα τέσσερα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στα διάφορα εργαστήρια ε, τις των σεμιναρίων πρώτα το μέλλον των σχέσεων Αφρικής Ευρωπαϊκής Ενώσεως Όσον αφορά αυτό το θέμα, υπογραμμίσαμε ότι η Ευρώπη και η Αφρική θα κερδίσουν εκεί οι δύο μέσω της ενισχύσεως των δεσμών τους. Θα πρέπει όμως να υπάρχει καλύτερο συντονισμό στις διάφορες δράσεις, στα διάφορα ζητήματα που γνωρίζετε. Εξίσου καλά εσείς όπως και εγώ και καλύτερα από μένα. Αλλά τα μεταστατικά φαινόμενα, η καταπολέμηση τρομοκρατίας, η αλλαγή του κλίματος, η διατήρηση της ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων και θα προσέθετα και η αρμονική ανάπτυξη της Γεωργίας την πρώτη συζήτηση της Συγκρατώ. ότι οι Οικονομική και Κοινωνική κοινωνικοί φορείς της Αφρικής θα πρέπει να είναι συνομιλητές μόνιμοι των πολιτικών φορέων και ανάντι και κατάντι ε, του καθορισμού στρατηγικών και αυτό συνεπάγεται επίσης ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της χρηματοδοτήσεως για τους προσώπους ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών. Κάτι που δεν είναι αυτονόητο αν θέλουμε να υπάρχει σωστή ε, ολοκλήρωση των αποστολών. Περισσότερη παιδεία και αύξηση εκπαίδευση και τον αύξηση των δεξιοτήτων κυρίως των νέων. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενώς, αλλά θα περιοριστώ να πω ότι είναι σαφές ότι το πρόβλημα της νεολαίας στην Αφρική όλος ιδιαίτερος είναι το πρόβλημα που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα θεματολόγια και εκεί θα πρέπει να τους δώσουμε λόγο στους νέους και στους προσώπους των νέων ούτως ώστε να μπορέσουν να παρουσιάσουν το όραμά τους, τις προσδοκίες τους όσον αφορά ε, την κοινωνία και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται διότι εκείνη πρωτίστως είναι το μέλλον αυτής της ε, Υπήρου. Αναφερθήκαμε στην ανάγκη ε, καθολική για όλους ε, και να υπάρχει μια συντονισμό εκπαιδεύσεω και αγορά εργασία και θα πρέπει να είναι εύκολη χρηματοδότηση των νέων σε περίπτωση ε, που θέλουν να φτιάξουν μια επιχείρηση. Μετά, μετά συζητήσαμε τη σημασία που έχει η γεωργία και ο αγροτροφημικός τομέας για να μεταμορφωθεί η Αφρική. Ε, υπενθυμίστηκε ότι αυτό που είναι θεμελιώδες και επίσης για την νεολαία και για να θετήσει να μην φεύγουν από την ύπεθρο είναι να γίνει Ήπεθρος ελκυστική, να μην φεύγουν οι νέοι, να μην ε, ερημώνεται η Ήπεθρος. Θέλουμε να δημιουργηθεί θετικός φαύλος κύκλος μέσω δημιουργίας διαφόρων επιχειρήσεων θετικών, ε, να δημιουργηθούν υποδομές, να ενισχυθεί κατάρτιση, ολοκλήρωση περιφερειακή, ε, χρειάζεται πίσω στους προπολογισμού. Όταν μιλάμε για τις διάφορες πολιτικές, υπάρχει ανάγκη να υπάρχει συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Δεύτερο σημείο το οποίο προβλήθηκε και ένας από τους βουλευτές το ανέφερε τώρα και πιστεύουμε πολύ σε αυτό που αναφέρθηκε είναι να προθίσουμε ε, τα παραδείγματα, την αξία των παραδειγμάτων μέσω της πολιτικής διαδόσεως έργων και προγραμμάτων που πέτυχα σε διάφορες χώρες Αφρικής θα το πετύχουμε αυτό. Δεν, δεν μιλάμε αρκετά γι' αυτό και έχουν υλοποιηθεί όμορφα πράγματα σε κάποιες χώρες, καλά πράγματα και είναι κρίμα που αυτά τα καλά επιτεύγματα δεν είναι τόσο ευρέως γνωστά. Θα πρέπει να εντοπιστούν και υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό. Ένας φορέας όπω το ΦΑΟ ε, που επεξεργάζεται την σπατάλη των τροφίμων μπορεί να διαδώσει τις καλές πρακτικές, να τις γνωστοποιεί. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, άμα δίνετε 15 δευτερόλεπτα ακόμα να πω ότι το τέταρτο σημείο που θέλω να αναφέρω συζητήθηκε με την κοινωνία των πολιτών της Αφρικής και της Ευρώπης είναι η ανάπτυξη της πράσινης ε, ενέργειας. Ε, η μετάβαση ενεργειακή είναι μια μέρημνα και ανησυχία μεγάλη, διότι μπορεί να οδηγήσει και σε οικονομική ανάπτυξη και θέση απασχόλησης στην Αφρικανική Ήπειρο. Το πάνελ μας ε, αναφέρθηκε σε ένα έργο που αναπτύχθηκε στην Ήπεθρο ε, της ακτής του ελεφαντοστού. Το εξετάσαμε αυτό. Ε, πρόσβαση ηλεκτροδότηση της υπαίθρου εφαρμόστηκε και πραγματικά ευαισθητοποιήθηκε και ο ντόπιο πληθυσμό όσον αφορά να υπάρχει τελικά μια απόσβεση του έργου και τελικά να ξεφύγουν από τη σχέση ε, δανειολήπτη-δανειοδότη. Και βρίσκουμε ότι το σύστημα βαθμολόγηση, το benchmarking, θα έπρεπε να αναπτυχθεί εκεί για να μπορέσουν να διαδοθούν οι καλέ πρακτικέ που εφαρμόζονται. Υπάρχει το παράδειγμα το συγκεκριμένο στην ε, περιοχή τη Ακτή Ολεφόντα του, αλλά και ε, μία κοινοβουλευτική συνέλευση εδώ και ένα χρόνο Στη Σομερή, στην Ναμίμπια συνέλευση, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο του Βινχουκ και, και είδανε τι γίνεται με ηλιακούς φούρνους που εκεί χρειάζονται λίγα σχετικά χρήματα αλλά επιτρέπουν τη δημιουργία θέσης απασχόλησης στην Ήπεθρο. και αυτό το παράδειγμα θα μπορούσε να προβληθεί περισσότερο. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά κυρία Πρόεδρε που μας ε, βοηθήσατε να διαφωτίσουμε, να μεταδώσουμε τα, αυτά που συζητήθηκαν στο Αμπιτζάν που οδήγησε τελική δήλωση. Ε, δήλωση που την αποστήλαμε στους διάφορους πολιτικούς υπεύθυνους. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ να μοιραστείτε μαζί μας τις εμπειρίες σας. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε τους κοινωνικούς εταίρους αυτά που συζητάμε. Σημαντική συνεισφορά. Να πω μερικά λόγια κι εγώ. Εγώ ήμουν επικεφαλής αντιπροσωπής επιτροπής μας και συμφωνούμε με αυτά που υπόθηκαν συναδέλφους. Πάντα λέμε ότι είναι σημαντική η ηγεσία στις χώρες. Καλός ηγέτης και καλά συστήματα διακυβέρνησης κάνουν τη διαφορά θέλουμε να δαπανώνται καλά τα χρήματα της βοηθείας μας και ότι βελτιώνεται η ζωή των διαφόρων λαών στις χώρες τους. Ε, δημιουργείται το αίσθημα πρόσφατα ότι υπάρχει μια νέα γενιά ηγετών, Αφρικανών ηγετών που αναδύεται, που θέλει διαφορετική προσέγγιση για το μέλλον. Μίλησα με νέους βουλευτές της ακτής του Ελεφαντοστού. Η Σεσίλ αναφέρθηκε σε εκπροσώπους της Γκάμπια, είχαμε εκπροσώπους του Κοινοβουλίου της Νιγηρίας και η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής πτυχής είναι σημαντικό κομμάτι της προσπαθίας. Ήμουν, ήμουν παρούσα στη διακήρυξη του Αμπιτζάν. Δεν ξέρω, θα βρει ε, θα ενταχθεί στη νέα κοινή στρατηγική που αναπτύσσετε εσείς. Διότι, αν σκεφτείτε το θέμα, ξέρουμε ποια είναι η ευρωπαϊκή εμπειρία. Μόνο όταν αυξήσαμε τη δημοκρατία είχαμε καλύτερη διακυβέρνηση. Δίνει αποτελέσματα για το λαό. Η λογοδοσία, ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για οικονομική ανάπτυξη. Και πιο δίκαιο επιμερισμό του πλούτου. Όταν ήμασταν εκεί, έγινε και μια ειδική συνάντηση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Υποτιμούμε την τοπική αυτοδιοίκηση στην οικονομική ανάπτυξη. Εγώ εργαζόμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα έπρεπε να το πω αυτό. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κοντά στον κόσμο. Μπορεί να κάνει την πραγματική αλλαγή φθηνά και γρήγορα. άκουσα τη Σεσίλ. Εμείς έχουμε μια εικόνα για προγραμματισμό, επενδυτικά προγράμματα. Το είπε και ο Σαλ. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας. Μεγάλα έργα από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες μεγάλες εθνι... Ε, πολυεθνικές ΜΚΟ και έχουμε οικονομική στήριξη, αλλά δεν έχουμε αρκετά μικρά έργα τα οποία θα μπορούσαν να στηρίξουν επιτόπου μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε τέτοια έργα και προγράμματα στη δική μας περιφερειακή πολιτική. Εγώ εργαζόμουν στην περιφερειακή πολιτική όταν ήμουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν στην πρώτη γραμμή εκεί. Προσπαθούσε να στηρίξει τον κόσμο επιτόπου, στη βάση. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να φανταστεί κανείς ένα ταμείο ε, ε, για βιώσιμη ανάπτυξη να, να, να χρηματοδοτήσουμε μικρά ποσά κάποια μικρά προγράμματα. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε πολλές μικρές μονάδες που χρηματοδοτούνται με μικρά ποσά, εφαρμόζουν έργα, δίνεται τεχνική βοήθεια σε, σε μικρή κλίμακα, να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις, να δούμε τι γίνεται στη Γενική Διεύθυνση για τις Περιφέρειες, τι γίνεται στις χώρες μας λίγο παραπάνω, πώς οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν, πώς μπορεί να τις στηρίξεις. Καινοτόμες ιδέες θέλουμε. Να δούμε τι έχει αποτελέσματα στις χώρες μας και αυτές να χρησιμοποιήσουμε και να τις ανταλλάξουμε. Όταν ήμασταν εκεί, η Σύνοδος Κορυφής εσκιάστηκε από το σκάνδαλο της Λιβύης. Αυτό το θέμα με τους πρόσφυγες δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα κρούση στο Task Force και ελπίζω να μάθουμε τελικά τι γίνεται εκεί πέρα. Διότι αυτό έχει αντίκτυπο στη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική, αλλά και στις χώρες μας. Είναι αυτό για το οποίο δεχόμεθα περισσότερες επιστολές από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο. Μα ζητάνε από εμά να τους πούμε, ε, σαν ευρωβουλευτές, γιατί υποστηρίζετε αυτά τα προγράμματα όταν βλέπουμε ότι πολλούνται σαν σκλάβοι οι Αφρικανοί πολλούνται στις αγορέ στη Λιβύη. Και πώ εμπλέκεται σε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακούν από τα διεθνή ΜΜΕ και θέλουν να ξέρουν ε, ε, εμεί τι κάνουμε για όλα αυτά. Και πώ είμαστε ανακατεμένοι σε αυτά. Υπήρξαν και κάποια άλλα θέματα που ανεδίσαμε που πρέπει να εξετάσουμε. Επισκεφτήκαμε την μπανανοφυτεία και φαινόταν καλό το πρόγραμμα. Αλλά τι δυσκολίες αντιμετωπίζει το πρόγραμμα. Διότι ε, τα συνοδευτικά μέτρα έχουν σταματήσει. Λοιπόν, αφού είχαμε μια επιτυχία σε αυτό το έργο, δεν πρέπει να το λησμονήσουμε. να μην χαθεί η επένδυση σε, αυτούς, τους, σε αυτές τις χώρες για αυτά τα θέματα. Και όσον αφορά για τις τοπικές ε, ΜΚΟ, στην ακτή του ελεφάντος του ε, υπήρξε ένα αίτημα που ακούσαμε, μας ζήτησαν στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περίοδου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ενδεικτικά προγράμματα για την αρχή του ελεφαντοστού για που βελτιώνει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το φροντίζουμε περισσότερο αν θέλουμε να πετύχουν στόχους τους βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό να εμπλακεί περισσότερο κοινό των πολιτών και αυτά τα προγράμματα να έχουν διαφάνεια. Πάρα πολλέ φορέ είχαμε συνομιλητέ σε διάφορε χώρε όλων των κόσμων που δεν ξέρανε ακριβώ γιατί έχουν εμπλακεί στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλέ ήταν οι ερωτήσει και αν μπορείτε με συντομία να απαντήσετε. να πεισείς στα υπόλοιπα για το πώς σκοτώνουμε, αλλά ε, Φερβάγε, αλλά για να δούμε τις ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα το θέμα της κοινωνίας των πολιτών και τη συμμετοχή της όπως και εσείς. Και εμείς θεωρούμε ότι δυστυχώς δεν μπορούσε να ακουστεί η φωνή της τη δεύτερη μέρα που συζητάμε για την διακυβέρνηση. Ο, όμως ε, το θέμα ήταν οργανωτικό. Ήταν χαοτική αυτή η δεύτερη μέρα. Είχαμε δύο συμπρόεδρους και είπε ο πρόεδρος Κόντε ότι επειδή πιέζει ο χρόνος μόνο οι επικεφαλής κρατών μπορούν να μιλήσουν. Ε, αυτό προκάλεσε αγανάκτηση στην αίθουσα και άρα δεν μπόρεσε οι εκπρόσωποι της να λάβουν το λόγο. Πάντως ε, κατά τα άλλα Όλοι τον λόγο, κοινοβούλια, ε, επιχειρηματίε. Επομένω δεν είναι γενικευμένο αυτό το πρόβλημα, δεν είναι κανόνα το πρόβλημα για την κοινωνία. Και όταν συζητήσαμε το πρόγραμμα, συναντήσαμε επισήμους, η Μογκυρίνη συνάντησε υπουργού πριν την συνάντηση κορυφής και είπαμε ότι θα δώσουμε αγώνα να καλυφθεί η κοινωνία από το πρόγραμμα. Θα επιμείνουμε και θα το καταφέρουμε δεύτερον. Σαν τη διασπορά. Τα είπε η κυρία Κέγγε. Ε, βέβαια, θα πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερο και στα πλαίσια της μετώπισης του μεταναστευτικού επίσης θα το προσέξουμε. Τόσο αυτό το πρόγραμμα δράσης, την πολιτική διακήρυξη, ε, για τη διακήρυξη. Αυτά γίνανε σε αυτή την χαοτική καταληκτική ημέρα της ε, συνάντησης κορυφής και υπήρχε μια σύγχυση σε σχέση με το ποιο κείμενο τελικά εγκρίθηκε. Και ακολούθησε ανταλλαγή εντυπώσεων μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης και Ξελών μέχρι να καταλήξουμε στο τι αποδέχονται οι δύο πλευρέ. Το κρίσιμο ήταν εκείνη η παράγωση για το μεταναστευτικό. Και τελικά όμω το θέμα ξεκαθαρίστηκε. Να, γιατί πήρε χρόνο μέχρι ότου ενημερώσουμε εσά. Τώρα το πρόγραμμα δράση. Αυτό είναι συνδυασμό ουσία και χρονικών συνδικών. Δεν μπορούσαμε να το κλείσουμε στο Αμπιτζάν αλλά υπήρχαν αποκλήσεις απόψεων και έτσι δεν εξετάστηκε ενδελεχώς το θέμα των επενδύσεων. Και επειδή έχουμε όλα αυτά τα έργα που έχουν σχέση με τις επενδύσεις, οπότε και μείναμε στην διακήρυξη και είπαμε ότι σε τρεις που δεν είναι και πολύ να έχουμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα. Αυτό τώρα είναι η επόμενη φάση. Τώρα από πλευράς ουσίας τα θέματα τα πολιτικά. Κύριε Γιώργος και για σας το λέω αυτό και για άλλους εδώ γιατί πρώτα πρώτα από δικής μας πλευράς δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το κοινό ενδιαφέρον, συμφέρον δεν μιλώ τώρα για το εμπόριο, γιατί η συνάντηση κορυφής μας βοήθησε να αποκτήσουμε μια επίγνωση του τι θέλουμε. Ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, των επενδύσεων για την απασχόληση. Και αυτά τονίστηκαν και στην πολιτική δήλωση διακήρυξη. Αυτό όμως γίνεται με τη φύλαξη των όλων, όλων όσων κάνουμε. Ε, πάντα παραμένει η προσέγγιση μα σφαιρική, γενική, πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη τη διάσταση διακυβέρνηση, της δημοκρατίας, της οικονομίας, το πώς δεν θα αφήσουμε κανέναν απ' έξω, πώς θα καλυφθεί και η καταπονήση της διαφθοράς, όλα αυτά τα οποία αναφέρονται ή στην διακήρυξη, αλλά είναι αλήθεια, στην ε, ανακοίνηση οι επενδύσει και ο ιδιωτικό τομέα ετονίστηκαν γιατί πρόκειται για μια νέα διάσταση που θέλαμε να προσθέσουμε στην εταιρική μα σχέση. Τώρα για τα θέματα τη ασφάλεια. Σε τέτοιε συνδύσεις κορυφή τουλάχιστον στην Ολομέλεια δεν υπάρχουν τα περιθώρια για να καλύψουμε και άλλα θέματα. Αλλά και εδώ ήταν το θέμα των κοινών ενδιαφερόντων που δεν ήταν μόνο το Σαχέλ και η συμφωνία θέλαμε να καλύψουμε και άλλες περιοχές. Είναι θέμα ελληνικής, ανθρώπινης ελληνικής. Η προστασία. Πολύ σημαντικά για την Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θέλουμε να βαθμιστεί συνεργασία μεταξύ Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης για αυτά. Με αυτό το μνημονίο κατανόησης το οποίο προωθήσαμε και που θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Οπότε ήταν θέμα συμπληρωματικότητα, ήταν θέμα να αναλάβει τις ευθύνες της Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή την κρίση. Οπότε έτσι με δυναμικό τρόπο και με την συμμετοχή του Μουσαφάκη, του Κουτιέρες, σε Μογκερίνη, ε, υπήρξε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για την ε, ασφάλεια, συνεργασία, συνεννόηση. Γιατί τη συνεννόηση δεν υπάρχει κοινή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την μεταρρύθμιση, την τροποποίηση των κανόνων για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Όμως τώρα μιλάμε για την παγκόσμια διακυβέρνηση Οπότε με αφιτηρία των Πιτζάν έχουμε καλύτερη συνεννόηση και για τα θέματα των μεταρρυθμίσεων για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Που για την παγκόσμια διακυβέρνηση πρόκειται για τη μεταρρύθμιση των διεθνών χρηματοοικονομικών θεσμών. Οπότε αργά γρήγορα και αυτό το θέμα θα μπει στο θεματολόγιο, στην μέρη διάδειξη συζήτησε. Τώρα δύο λογάκια για τα συμπεράσματά σα, ε, Λίντα. Όσον αφορά την τοπική διακυβέρνηση, συμφωνώ 100% και για αυτό το λόγο. Και φέτο θα ξανασυζητηθεί αυτό. Πέραν τη κεντροκατευθυνόμενη διοίκηση, θέλω να δούμε τι γίνεται και στο τοπικό επίπεδο, πιο κοντά μέσα στον κόσμο. Σε άντρε και γυναίκε, Ακριβώς το θέμα της ηγεσία είναι πολύ σημαντικό και κατακλείδη αν κανείς ρίξει μια ματιά στα τσινά της θα δούμε ότι υπάρχει δυναμική ηγεσία τώρα ότι έχουν γίνει αλλαγές σε πολλές ε, χώρες και υπάρχει και το δημογραφικό άλλωστε οπότε και πολλοί αφορικανοί ηγέτες θα συνειδητοποιήσουν σύντομα ότι ήρθε η ώρα της αλλαγής αλλιώς δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτό τους όλους τους μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα στην Αφρική. Και ευχαριστώ. Κουν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν θα σχολιάζω διάφορα οργανωτικά θέματα για μια αποστολή που δεν οργανώσαμε εμείς. Να ξεκινήσω με το σχόλιο του κυρίου Γκέρενς για τις ιστεροβουλίες κάποιων κρατών μελών μας. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να εκτιμήσει κανείς τις ιστεροβουλίες γιατί δεν εκφράζονται. Το βασικό στοιχείο για μένα είναι ότι ανάμεσα στην ε, χρηστική προσέγγιση και τους στόχους της ανάπτυξης δεν υπάρχει αντίφαση. Αυτό θα πρέπει να τονίσουμε και να εξηγήσουμε ιδιαίτερα σε όσους για λόγους ε, ε περιορισμένης αντιμετώπισης δεν βλέπουν τη σύνδεση. Η Ευρώπη αντίθετα με άλλους δεν μπορεί να θεωρεί ότι μπορεί να πάει στην Αφρική να πάρει κάτι, να φύγει κλείνοντα την πόρτα και ε, να θεωρήσει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Γιατί αν έχουμε τέτοια προσέγγιση έναντι της Αφρικής, η Αφρική θα πάει χάλια και όταν πηγαίνει χάλια η Αφρική, αυτό έχει επιπτώσεις σε εμάς. Άρα, άρα από πλευράς ε, αν το δούμε. Είναι προς το ε, βασικό συμφέρον να έχουμε άλλη προσέγγιση προς αυτήν την Ήπειρο και όχι μόνο να μας ενδιαφέρει το βραχυπρόθεσμο περιορισμένο όφελος. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη συζήτηση δεν πρέπει να αποφύγουμε. Είτε για τα θέματα της μετανάστευσης, είτε για την οικονομική ανάπτυξη, είτε για θέματα ειρήνης και ασφάλειας. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτά τα θέματα, τότε απευθείας περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι ακριβώς η διακυβέρνηση, η βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η αντιμετώπιση της φτώχειας, της μείωσης των ανισοτήτων. Η Ευρώπη δεν θα εξυπηρετήσει τα άμεσα συμφέροντά της αν δεν έχει μια πιο ευρύτερη προσέγγιση. Αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το εξηγούμε, να το τονίζουμε και να το έχουμε ε, ως πηξίδα μας. Τώρα για το EIP. Πρέπει να τονίσουμε τα πάντα. Το EIP δεν είναι κάτι που βοηθάει τις πολυεθνικές. Ένα από τα βασικά κριτήρια ε, ένα, μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να χορηγηθεί ενίσχυση από το EFSD είναι να εγγυηθούμε την ε, ε, επιλεξιμότητα. Στην περίπτωση των πολυεθνικών και των μεγάλων επενδυτών η παρέμβασή μας δεν χρειάζεται. Δεν αλλάζει την κατάσταση. Άρα δεν το κάνουμε. Να προσθέσω κάτι άλλο. Ένα από τα παραθά, ένα παράθυρο που ετοιμάζουμε τώρα αφορά τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνούμε με πολλά από αυτά που είπατε. Είναι ότι για να δημιουργηθεί η αναγκαία οικονομική δυναμική, να αξιοποιηθεί το οικονομικό δυναμικό της Αφρικής, ούτως ώστε να ξεφύγουν από τη φτώχεια, φτώχεια οι Αφρικανοί και ιδιαίτερα οι Αφρικανές, είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτήσει. Έχουν την επιχειρηματικότητα, έχουν το δυναμικό, δεν έχουν τους αναγκαίους πόρους ή αυτοί οι πόροι δεν φτάνουν στους απλούς πολίτες. Λοιπόν, ένας από τους στόχους για ε, την επίτευξη αυτού του στόχου, μάλλον ένα από τα μέσα για την επίτευξη του στόχου είναι η χορήγηση εγγυήσεων μέσω της διευκόλυνσης εγγυήσεις σε διάφορες ε, τράπεζες είναι όπως λειτουργεί το ΕΦΣΙ συνολικά. Δίνουμε εγγυήσει στις τράπεζες που θα επιτρέψει στις τοπικές τράπεζες που συνομιλούν με τους πολίτες δεν είναι ε, η ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή η, τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Τράπεζα συνεργάζονται με τοπικές τράπεζες και έτσι έρχεσαι σε επαφή με τους απλούς ε, επιχειρηματίες των χωρών αυτών. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Και συμφωνώ με αυτό που ανέφερε και ο κύριος Σονβίλ. Ε, η σημασία ορισμένων τομέων της οικονομίας και ιδιαίτερα του γεωργικού είναι πολύ βασική. Εκεί υπάρχει τεράστιο δυναμικό από μία, είναι ένας τομέας που απασχολεί ε, πολλούς Πολλοί βέβαια ε, ασκούν τη γεωργία σε επίπεδο απλό επιβίωσης αλλά έχουν περισσότερες δυνατότητε, έτσι δημιουργούνται αλυσίδες αξίες γίνεται η σύνδεση μεταξύ των μικρογεωργών με τις τοπικές αγορές και κατόπιν τις ε, πιο σημαντικές, πιο μεγάλες περιφερειακές ε, αγορές. Αυτή είναι μια δυνατότητα που ήδη αναπτύσσουμε και θέλουμε να προωθήσουμε περισσότερο επειδή όλα βέβαια αλληλοσυνδέονται. Η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα είμαι πολύ ε, σύντομος. Βεβαίως οι τοπικές αρχές είναι πάντα ε, προτιμησιακοί συνομιλητές μας. Σε επίπεδο πόλεων επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε πόλους αναπτυξιακούς. Λοιπόν, επειδή πρέπει να ολοκληρώσω, για την μετακοτονού εποχή. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, γιατί αύριο πρωί θα έχετε τη δυνατότητα να το συζητήσετε, αν δεν κάνω λάθος, με τον Επίτροπο Μίμητσα, τον ίδιο. Λοιπόν, να πω μόνο ότι έχουμε εδώ τον τετραγωνισμό του κύκλου μεταξύ της μετακοτονού εποχής με τη Βόρεια Αφρική και την Ποσαχάρη Αφρική μέσω της ε, Αφρικανικής Ένωσης, νομίζω ότι επετεύχθη αυτός ο τετραγωνισμός. Στις ε, κατευθύντριες ε, διαπραγματευτικές γραμμές που εγκρίναμε και τώρα συζητάμε με τα κράτη-μέλη, εξηγούνται όλα αυτά και είναι σαφές ότι εφόσον θέλουμε να συνομιλήσουμε με την Αφρική για το μέλλον της Αφρικής, μετά το Κοτονού ακριβώς πρέπει να συζητήσουμε με την υποσαχάρια Αφρική αλλά όχι μόνο, με ολόκληρη την Αφρική πώς ακριβώς θα συμβεί δεν έχω χρόνο τώρα να σας εξηγήσω, αλλά ε, διατυπώνεται σαφώ την πρότασή μα αυτή σε αυτό το κείμενο των διαπραγματευτικών κατευθυντηρίων γραμμών και αν θέλετε θα τα συζητήσουμε αργότερα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε για την μετακοτονού εποχή. Θα γίνει ένα ειδικό εργαστήρι, workshop γι' αυτό. Θα έχουμε πολύ χρόνο για αυτή την περίοδο. Ευχαριστούμε του ε, δύο μιλητέ. Πολύ ωραία επισκόπηση και παρακαλώ να μας ε, τηρείτε ε, νήμερους για αυτή την κατάσταση. Σας παρακαλώ ε, όλοι εκτός από τους συντονιστές και όσους επιτρέπετε να μείνουν εδώ να αποχωρήσουν αύριο στις 9. Σας υπενθυμίζω ότι είστε όλοι προσκεκλημένοι στις 6.30. Στις 6.30 λέω. 6.30 λέω. Όπως είπα το πρωί ή αν αποχωρεί και θα κάνουμε μια δεξίωση για να ε, την ευχαριστήσουμε. Χαίρετε.